από τη συντονίστρια, μια συντονίστρια ακούσαμε ότι βρίσκεται ε, καθοδόν, έχει πρόβλημα στην κυκλοφορία, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο, είναι 9 και 4 σχεδόν. Θα ήθελα να καθίσετε όλοι να ξεκινήσουμε. Έχουμε την σε συγκρότηση συνεδρίασή μας, ε, συντακτική σε συγκρότηση της Επιτροπής μας και Έχουμε και ε, στόχο να εκλέξουμε το νέο πρόεδρο και τους νέους αντιπροέδρους για την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα έχουμε την απαρτία, χρειάζονται μόνο 13 για απαρτία για τις εκλογές αυτές μετά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ευτυχώς ή δυστυχώς έχουμε τον κανονισμό, δηλαδή το άρθρο 12 του κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου, ότι ο προηγούμενος πρόεδρος θα προεδρεύει για την εκλογή του επομένου πρόεδρου. Έχουμε την κατάσταση αυτή. Εγώ θα προεδρεύσω λοιπόν κατά την εκλογή του νέου ή της νέας πρόεδρου. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να δείξετε κατανόηση δεν θέλουμε, παρα, να, δεν θέλουμε να παραβιαστεί ο κανονισμός, γι' αυτό γίνεται αυτό. Ξεκινάμε με την εκλογή Προέδρου. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι Λάμπερτ Φανίστερ Ρόι, εξ ονόματος του ΕΛΚΑ. Έχετε τον λόγο κύριε Φανίστερ Ρόι. Σας ευχαριστώ πολύ δεν θα έπρεπε να σας κρατήσουμε επί μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτή τη δύσκολη θέση να προεδρεύετε. Το επεξηγήσατε. Δύσκολο είναι να κατανοήσει κανείς ε, το πώς αισθάνεται κάποιος. Είναι όμως ε, τιμή και χαρά πρέπει να πω ότι το ΕΛΚ επιθυμεί να προτείνει την κυρία Χιμπνερ, Ντανούτα Χούμνερ ως ε, υποψήφια επόμενη πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής και θα έχει και καλύτερες επιδόσεις από ό,τι και στο παρελθόν. Πράγμα πολύ δύσκολο, ανέφικτο ίσως. Όμως υποψήφια του ΕΛΚΑ για το δεύτερο ήμιση αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας ως πρόεδρος, η κυρία Ντανούτα Χιούμπνερ λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχα την υποψία αυτή. Γι' αυτό είπα ότι ήμουν αμήχανη, αισθανόμουν μεγάλη αμηχανία να προεδρεύω. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, πρέπει να πω ότι ναι, αλλά πρέπει να το πω ότι συμφωνώ εγώ να είμαι υποψήφια. Είναι σημαντικό και αυτό, έτσι. Ο κύριος Φανίστερ Ρόι πάλι, παρακαλώ. Μάλιστα. Ίσως επειδή σε σχέση με τα μέλη της Επιτροπής για την εκλογή, ίσως αν άλλος υποψήφιος δεν υπάρχει διαβοής, μπορείτε να εκλεγείτε τώρα. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια λέει ο κύριος Φανίστερ Ρόι. Η κυρία Χίμνε, σας ευχαριστώ πολύ να σας δώσω άλλη μια πληροφορία ότι σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί η δήλωση οικονομικών συμφερόντων από πλευρά μου. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ για αυτό που κάνατε και ελπίζω ότι το δεύτερο ήμιση της κοινοβουλευτικής μας θητείας, της νομοθετικής θητείας που θα αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το τι θα πρέπει να κάνουμε, με χαρά θα στραφούμε στο έργο και μεγάλη ικανοποίηση αλλά υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να προχωρήσω στο δεύτερο σημείο αυτή τη συγκρότηση της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής, επιτροπή ε, εκλογή των αντιπροέδρων. Έχουμε το δικαίωμα να έχουμε μέχρι τέσσερις ε, αντιπροέδρους. Στο σημείο τρία η εκλογή των αντιπροέδρων για το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Η διαδικασία ουσιαστικά είναι πάλι ίδια. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εσάς τους συντονιστές ποιες είναι οι προτάσεις σας για υποψηφίους. Έχουμε τέσσερις αντιπροέδρους που ας το πω έτσι έχουν αξιωματικά τη θέση τους ε, γύρω από την πρόεδρο. Πρώτος αντιπρόεδρος, δεύτερος αντιπρόεδρος, τρίτος, τέταρτος αντιπρόεδρος και θα πρέπει να συμφωνηθεί επίσης ε, από πλευρά τους να είναι υποψήφοι και θα πρέπει να επικυρωθεί ότι έχουν όπως πρέπει συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων από πλευράς τους και την έχουν καταθέσει. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την Κωνσταντσε Κρέλ. Αναζητούμε υποψήφιο ή υποψήφια για τον πρώτο αντιπρόεδρο ως αξίωμα. Σα ευχαριστώ πολύ. Πρώτα συγχαρητήρια σε εσά, Ντανούτα, για την επανεκλογή σα. Θέλω να προτείνω εξ ονόματο των Σοσιαδημοκρατών τον κύριο Σταυρακάκη ω πρώτο πρόεδρο. Εξαιρετική δουλειά έκανε κατά τα τελευταία δυόμιση χρόνια ο κύριο Σταυρακάκη. Είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνει και εξαιρετική δουλειά κατά τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Η κυρία ε, Ντανούτα Χιούμπνερ, να ρωτήσω, υπάρχουν άλλοι υποψήφοι ως ε, πρώτος, για το αξίωμα του πρώτου αντιπροέδρου τη Επιτροπή μα, Αν όχι, Κύριε Σταυρακάκη, εσείς θα πρέπει να μας πείτε ότι δέχεστε αυτή την πρόταση και έχετε συμπληρώσει το, τη δήλωση. Thank you very much, ε, Σας ευχαριστώ πολύ Ντανούτα. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Ευχαριστώ τη συντονίστρια και τους συναδέλφους μου για αυτή την πρόταση. Να είμαι υποψήφιος, δέχομαι αυτή την πρόταση με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ. Η κυρία Χρύμπνε, πρόεδρο. Τώρα να ρωτήσω τον κύριο Λάμπερ Φανίστερ Ρόι. Πρόταση για τον δεύτερο αντιπρόεδρο, την δεύτερη αντιπρόεδρο ο κύριος Φανίστερο. Υποψήφιος για μας θα είναι ο Μάρκο Πίπερ υποψήφιος για το αξίωμα του Δευτέρου Αντιπροέδρου αυτής της κοινοβουλευτική μα επιτροπής. Αυτή είναι η πρότασή μα από το ΕΛΚ. Η κυρία Χίβνερ. Φαίνεται να έχει εκπλαγεί ο Μάρκο. <laughs> Ελπίζω ότι συμφωνείτε Μάρκο. Συμφωνείτε. Όλο και περισσότερο φαίνεται ότι κάτι με εκπλήσει, αλλά με ιδιαίτερη χαρά το δέχομαι. Ευχαριστώ. Η κυρία Χίμπνε, πρόεδρο. Οι συνάδελφοι υποθέτω ότι έχουν συμπληρώσει τι δηλώσει οικονομικών συμφερόντων από πλευρά του και τώρα θα ήθελα να προχωρήσω και να ζητήσω υποψήφιο για τον τρίτο αντιπρόεδρο το πρόβλημα είναι ότι... Α, εντάξει, εσείς θα θέλατε να μας ενημερώσετε εξ ονόματος των φιλελευθέρων την πρόταση για το αξίωμα του τρίτου αντιπροέδρου. Πρώτα απ' όλα, εξ ονόματος της Άντε, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια να εκφράσω τα συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Για τρίτο αντιπρόεδρο υποβάλλουμε την κυρία Ισμανόβα ως υποψήφια. Δεν παρίσταται. Όμως μπορώ να σας πω ότι δέχεται αυτή την πρόταση να εκλεγεί ως τρίτη αντιπρόεδρο. Δεν παρίσταται. Αλλά από ό,τι μας είπατε συμφωνεί, έτσι. Εντάξει, σας, ε, σας ευχαριστώ να ρωτήσω ε, εσείς τώρα για τον υποψήφιο των Πρασίνων. Τι προτείνετε. Euh, Θα ήθελα να σας συγχαρώ κυρία Πρόεδρε και να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας ε, που ανανεώθηκε. Έχουμε ε, τον συνάδελφο Τρεμόπουλο που είναι υποψήφιος για τη θέση του τετάρτου αντιπρόεδρου. Ευχαριστώ. Η κυρία Χίμνερ, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Τρεμόπουλε, συμφωνείτε με αυτή την υποψηφιότητα όπως προτάθηκε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ για την τιμή, συγχαρητήρια και εσάς. Καλή συνέχεια. Thank you. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τρεμόπουλε. Δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι από ό,τι βλέπω που να, υπάρχουν, να υποβάλλονται από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Προτείνω λοιπόν, μια και έχουμε ακριβώς τον αριθμό των υποψηφίων που ανταποκρίνονται στα αξιώματα αντιπροέδρων που πρέπει να επανεκλεγούν, προτείνω να διαβοήσουν να εκλεγούν. Και αν θα μπορούσαμε ομού να ψηφίσουμε διαβοής. Δεν υπάρχει πρόβλημα και ομού και διαβοής. Ευχαριστώ. Um, uh, unfortunately, there is the first job to do. Τώρα, θα ήθελα να σας ζητήσω να έρθετε εδώ τώρα, οι εκλεγέντες αντιπρόεδροι, να καθίσετε δίπλα μου εδώ στο Προεδρείο. Αυτό λέει ο κανόνισμος. So, dear colleagues, uh, could you please join me here? Uh, Λάτε να καθίσετε εδώ, κοντά μου στο Προεδρείο. Thanks. Λυπούμε. Είχα συγκινηθεί και δεν ε, σας συνεχάριν πιο πριν. Θέλω να σας συγχαρώ και τους τέσσερις σας για την εκλογή σας αυτή. Και τώρα θα ήθελα να κλείσουμε αυτή τη συνεδρίαση σε αυτή τη στη φάση. Από ό,τι γνωρίζω έχουμε και συντονιστές που εκλέγονται, ε, έχουν επανεκλεγεί. Τώρα όλα είναι στη θέση τους, όλοι είναι στα αξιώματά τους, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σκληρή δουλειά που μας περιμένει. Να ξεκινήσουμε τώρα λοιπόν, μετά από αυτό, να ξεκινήσουμε με την τακτική μας συνεδρίαση, που ως ήθιστε <clears throat> θα ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω στο σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή έγκριση της ημερήσιας διάταξης, ότι δεν είχαμε κάποιες προτάσεις. Για πρώτη φορά δεν υπάρχουν προτάσεις αλλαγής του σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν προτάσεις και τώρα για κάποια αλλαγή, θα ήθελα να πω ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Μάλιστα, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Και περνάμε αμέσως στη συνέχεια στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασής μας του Νοεμβρίου, 22ης και 23 η Νοεμβρίου 2011. Και όπως συνήθως είναι στη διάθεσή σας τα πρακτικά και έχουν διανεμηθεί και ως ήθιστε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρηθεί ότι επικυρώνονται εκτός αν υπάρξουν κάποιες ενστάσεις και αντιρρήσεις. Για το επόμενο σημείο στη συνέχεια στην ημερήσια διάταξη, ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν έχω κάποια ανακοίνωση να κάνω σε αυτή τη φάση. Οπότε μπορούμε αμέσως να περάσουμε στη συνέχεια στο επόμενο σημείο στη Μέση Διάταξη, που είναι ησυχία παρακαλώ. It's usual that assistants speak much more loudly than the... Λοιπόν, σε σχέση με τις φωνασκίες ε, ε, υπάρχει κάποια φασαρία θα πρέπει να σταματήσει αυτή γιατί αλλιώς πρέπει να μιλάμε πολύ δυνατά. Διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών τώρα. Η συγγήτρια η κυρία Εσμπέτα Καταζίνα Λουκασεύσκα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εδώ κάτι. Να υπενθυμίσω σε εσά το εξή. Κάποιοι ίσως δεν το έχουν ακούσει και γι' αυτό θέλω να ενημερώσω όσους δεν το έχουν μάθει. Για όσους δεν το έχουν πληροφορηθεί, να το πω λοιπόν, έχουμε κατεπήγοντα χαρακτήρα, ασυνήθιστη κατεπήγουσα κατάσταση. Είδαμε ότι η φωνή μας όσον αφορά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων πρέπει να εισακούγεται, διότι η ευρωπαϊκή πολιτική στη μεθοδολογία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων. Γι' αυτό Θέλαμε λοιπόν να γνωμοδοτήσουμε προ την ΕΚΟΝ, την ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών Θεμάτων, με αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλία. Και ζητώ λοιπόν σε σχέση με την ε, ψηφοφορία για την 5 και 6 Φεβρουαρίου ζήτησα από, με επιστολή από πλευράς ε, της Προεδρίας της ΕΚΟΝ να αναβληθεί και να ακολουθηθεί η κανονική τακτική διαδικασία στην κοινοβουλευτική μα επιτροπή. Αυτό όμω είναι αδύνατο, είναι ανέφικτο. Γι' αυτό πρότεινα στου συντονιστέ να εγκρίνουμε με αυτή την ασυνήθιστη διαδικασία, το οποίο σημαίνει ότι στις 15 Ιανουαρίου, με την αποστολή του σχεδίου έκθεσης σε εσά, ζητώντας σας να προετοιμαστείτε για ένα πολύ πιεστικό στενόχρονο διάγραμμα, με προθεσμία πιεστική για την κατάθεση τροπολογιών σήμερα δηλαδή μετά την ε, συζήτηση της ε, παρουσίασης και των σκέψεων του σχεδίου έκθεσης διότι πρέπει να ψηφιστεί και να εγκριθεί αύριο για να διευθετηθεί. Θέλω να σας το πω και να το συνειδητοποιήσουμε αυτό ότι θα εξετάσουμε αυτή την γνωμοδότηση προθεσμία για τροπολογίες θα ανοίξει μόνο μία τροπολογία λέγεται μόνο μία τροπολογία έχουμε μέσω αυτής της διαδικασίας επίσπευσης, ας το πω έτσι, εξέτασης τροπολογιών, μία τροπολογία, ε, προθεσμία μέχρι τις 4 το απόγευμα σήμερα, θα ψηφίσουμε αύριο. Αυτό είχε συμφωνηθεί με τη γραπτή αυτή διαδικασία, για αυτήν την ασυνήθιστη διαδικασία με τους συντονιστές. Δίνω τον λόγο στην κυρία Λουκασιεύσκα τώρα παρακαλώ. Εσμπιέτα παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους σας για τη συμφωνία σας με την ε, γρήγορη διαδικασία. Γιατί η διαδικασία, κυρίως όσον αφορά με αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα, είναι σημαντικά, είναι σημαντικότατες οι ευρωπαϊκές στατιστικές. Η Ρέτζι είναι μια πολύ σημαντική επιτροπή που πρέπει να έχει στη διάθεσή της ποιοτικά δεδομένα για να διαπιστώνει αν εκτελούνται όντως οι, αρχικές, οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές εάν προωθούνται στρατηγικές οι οποίες βοηθούν όντως την ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε κατά συνέπεια καλά στατιστικά δεδομένα που με τη σειρά τους θα μας βοηθήσουν να περιφρουρούμε καλύτερα τις φορολογικές και μακροοικονομικές πολιτικές. Εγώ επιστήνω την προσοχή σας στο πόσο είναι σημαντικό να σεβόμαστε την εμπιστευτικότητα των στοιχείων όταν μιλάμε για στατιστικές. Και αναρωτιέμαι αν αυτή η ενιοποίηση που προτείνει η ΕΚΟ σχετικά δηλαδή με το θέμα των δημοσίων λογαριασμών είναι θεμελιώδης. Θέτω αυτό το ερώτημα μέσα στα πλαίσια του κανονισμού, ο οποίος ε, ενημερώθηκε μετά από την ανακοίνωση της Κομισιόν σχετικά με τα όσα συνέβησαν στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι υπήρξε μία ε, επίσκεψη στην Ελλάδα για διαβουλεύσεις και μετά έγινε και μία επιθεώρηση για να βελτιωθεί ο έλεγχος των πηγών των δεδομένων. Κατά τη γνώμη μου στον κανονισμό τα κράτη-μέλη θέλησαν να ευθυγαρμιστούν με αυτήν την μεθοδολογία, η οποία βέβαια αυξάνει το κόστος. Χρειάζονται λοιπόν αποτελεσματικά μέτρα σήμερα που θα επιτρέψουν σε όλα τα κράτη-μέλη να λειτουργούν εύρυθμα. Επίσης, στη γνωμοδότησή μου επιστήνω την προσοχή στο γεγονός ότι χρειάζεται να επεξεργαστούμε ένα κοινό σύστημα έρευνας για τα στοιχεία που αφορούν την διερεύνηση κοινωνικο-οικονομικών στοιχείων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το σκέλος ανάπτυξη και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει εμείς από κοντά να βλέπουμε ποιες είναι οι κοινωνικο οικονομικές πραγματικότητες, στις διασυνοριακές περιοχές, στις αστικές περιοχές και στην Ήπεθρο. Χρειάζεται επίσης και μία μεθοδολογία που να αφορά στα σύνορα, με τις τρίτες χώρες και τα εσωτερικά σύνορα Σέγγεν. Χρειάζονται πιο αποτελεσματικά ερευνητικά συστήματα συστήματα για τα ισοζύγια πληρωμών και για την επαλήθευση, των έλεγχο των λογαριασμών περιφερειακών και εθνικών. Αυτό σημαίνει καλύτερη ποιότητα. Η Κωνσταντσα Κρέλ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια και πραγματικά μπορώ να πω κάτι το οποίο ίσως είναι ασυνήθιστο στο σώμα. Υποστηρίζουμε απόλυτα αυτό το οποίο μόλις μας εκθέσατε, αυτό το οποίο εμπεριέχεται στη γνωμοδότηση. Δεν θα θέσουμε τροπολογίες, δεν θα καταθέσουμε τροπολογίες. Ευχαριστώ πραγματικά για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ε, thank you. Ευχαριστώ. Η κυρία Μανέσκου. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Μανέσκου. Μάικρο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τη συγχαίρω. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να μπορεί κανείς να συντάξει ε, μια γνωμοδότηση. Η ομάδα ALDE συμφωνεί με το κείμενο και δεν πρόκειται να υποβάλει τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ε, ο Ζων Πολ είναι εδώ. Ο συνάδελφος από τους Πράσινους δεν είναι εδώ, αλλά έχουμε λάβει ε, τροπολογία από τους ε, πρασίνους. Δεν ξέρω μήπως ε, θέλετε να σχολιάσετε. Δεν υπάρχουν πολλά σχόλια που θα μπορούσαν να γίνουν απαντώντας στους σκιώδεις. Α, με συγχωρείτε. Υπάρχει ακόμα ο Λόμπερ. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό νομίζω. Στο σημείο 4 λέγεται για τις διασυνοριακές περιοχές και στο σχόλιο σας ε, λέτε επίσης ε, για τα εξωτερικά σύνορα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα διότι χρειαζόμαστε αυτές τις ε, πληροφορίες σχετικά με τα εσωτερικά σύνορα και με τα εξωτερικά σύνορα επίσης. Ίσως μπορούμε κάτι να προστάσουμε εδώ. Το έχετε περιλάβει αλλά ίσως δεν είναι στο κείμενο. Λέτε τα εξωτερικά σύνορα. Τα άκουσα στα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συντονιστές και θα λάβω υπόψη μου όλα όσα είπε ο κύριος Βανίστερόη και θα κοιτάξω να τροποποιήσω σχετικά το κείμενό μου. Για την τροπολογία των πρασίνων θεωρώ ότι πρέπει να απορριφθεί. Ευχαριστώ, ναι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ εκπροσωπώ εδώ τον κύριο Βεσέτ που είναι άρρωστος. Εμείς διατηρούμε την τροπολογία μας. Και θα μπορούσε να την δεχτεί κάλλιστα η συγγήτρια, διότι είναι μια τροπολογία με νόημα για ε, ε, σχετικά με τη συνοχή. Είναι μια τροπολογία η οποία τίνει να ε, ε, εντείνει την ίδια τη θέση της ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η μόνη απόφαση που λαμβάνουμε τώρα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες 4 το απόγευμα και θα ψηφίσουμε αύριο, αλλά έχουμε ακόμα χρόνο για συζήτηση ανάμεσα στους σκιώδεις και τις πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να κλείσουμε για αυτό το σημείο. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Τώρα έχουμε μια επιλογή διότι κανονικά ο κύριος Νίκολάι Βάμεν έρχεται σε μισή ώρα. Έχουμε τώρα μισή ώρα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για το σημείο της ημερήσιας διάταξης που βρίσκεται μετά την ανταλλαγή απόψεων με την Δανική Προεδρία, που είναι το σημείο για το οποίο εγώ είμαι υπεύθυνη. So we, I just explain to you what are the... Θα σας εξηγήσω ε, ποια είναι τα προβλήματα, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο για να αρχίσουμε τη συζήτηση για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Δεν έχουμε όμως εδώ το εκπρόσωπο της Επιτροπής ε, και της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων και της Greek Task Force. Αυτό νομίζω ότι είναι το αρνητικό, το κατά. Αλλά μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση χωρίς την παρουσία αυτών των εκπροσώπων. Σας ζητώ να αποφασίσετε. Ιδαλλιώς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διακόψουμε τη συνεδρίαση για αυτή τη μισή ώρα. Μέχρι τις 10. Μήπως οι συντονιστές έχουν κάποια γνώμη σχετικά με το θέμα αυτό. Έχω ε, νομίζω εγώ την δυνατότητα να αποφασίσω αν θα συνεχίσουμε ή θα διακόψουμε. Ε, όχι, ας αρχίσουμε λοιπόν. Το θέμα αυτό είναι αρκετά δύσκολο από την άποψη της διαδικασίας, διότι είναι ένα θέμα κατεπήγων, διότι πρόκειται για την τροποποίηση του κανονισμού που σκοπό έχει να διευκολύνει την πλήρη χρήση, η καλύτερη χρήση της χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμη για τα κράτη-μέλη σε σχέση με την ανάπτυξη, σε σχέση με τα πακέτα λιτότητα, σε σχέση με τα κονδύλια που υπάρχουν στο Ταμείο Σύνοχης και αυτό θα μπορούσε να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Η πρόκληση έγκυται στο γεγονός ότι το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμη αρχίσει να επεξεργάζονται το θέμα. Η ιδανική Προεδρία, ίσως ο Υπουργός Βάμεν θα μας ενημερώσει, αλλά μέχρι τώρα δεν υπήρχε κανένα χρονοδιάγραμμα, καμία ατζέντα, κανένα πρόγραμμα για το πώς το Ξυμβούλιο θα ασχοληθεί με αυτήν την τροποποίηση. Λόγω του κατεπήγοντος του θέματος, εδώ οι σκιώδεις και η συγγήτρια θα μπορούσαν να, να αρχίσουν μια ανάγνωση, αλλά αν κάνουμε μια ανάγνωση χρειαζόμαστε συνεργασία με τους ε, τρεις οργανισμούς κατά, κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μία μόνο ανάγνωση. Αυτό δεν είναι δυνατόν επειδή το Συμβούλιο σε αυτό το στάδιο δεν είναι σε στάδιο που θα μπορούσε να μας ε, ενημερώσει ακόμα και για την κατεύθυνση σχετικά με τον κανονισμό αυτό. Για μας λοιπόν η πρόκληση, αν θα αγνοήσουμε δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει κινητικότητα από πλευράς του Συμβουλίου και εμείς θα προχωρήσουμε με τη δουλειά μας και θα δούμε τι θα συμβεί όταν το Συμβούλιο αρχίσει τη δουλειά του ή αν ε, θα καθυστερήσουμε λίγο τη διαδικασία για να προσαρμοστούμε στην ταχύτητα εργασίας του Συμβουλίου και για να ασκήσουμε και κάποια πίεση στο Συμβούλιο είναι μια παράδοξη περίπτωση, διότι περιμένουμε τα πρώτα σημάδια, της πρώτες ενδείξεις κινητικότητας από πλευράς του Συμβουλίου. Εγώ προσωπικά σκέφτηκα ότι δεν έπρεπε ε, να κολλησιεργούμε και ότι θα πρέπει το Φεβρουάριο να έχουμε το σχέδιο εισήγησης της εισηγήτριας σας εξηγώ επίσης γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Θέλουμε να δράσουμε ταχύτατα και γι' αυτό περιμένουμε ορισμένες ενδείξεις, ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές από το Συμβούλιο που για την ώρα είχε μια συνεδρίαση το Δεκέμβριο που μόνο ερωτήσεις τέθηκαν στο τραπέζι, τέθηκαν στην Επιτροπή για επεξηγήσεις δεν υπήρχε καμία έκφραση των απόψεων που θα επικρατήσουν στο Συμβούλιο. Ε, γι' αυτό σας θέτω το θέμα για εξέταση, πρωτού περάσουμε στην ίδια την ουσία της συζήτησης αυτής. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι οργανώσαμε μια πολύ καλή τεχνική συνεδρίαση όπου οι περισσότεροι σκιώδεις εισηγητές συμμετείχαν με την ε, επιτροπή που εκπροσωπήθηκε όχι μόνο από την DG Regio αλλά ε, και από ε, την Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων που ήταν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό διότι αυτό το μέσο επιμερισμού του κινδύνου ε, δεν είναι κάτι το καινούριο, είναι κάτι το οποίο το έχει εξετάσει ε, για τα, τους άξονες ε, μεταφοράς, τα ευρωπαϊκά δίκτυα το έχει εξετάσει η Κομισιόν και για την περιφερειακή πολιτική. Ξέρετε το Jeremy είναι ένα μέσο παρόμοιο που υπάρχει και βοηθάει τις εταιρείες. Είχαμε λοιπόν ενδελεχή ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν και επίσης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που συμμετείχε σε όλες τις συζητήσεις μας και στην τεχνική συνεδρίαση όπου ήταν πάρα πολύ χρήσιμο διότι εξήγησε τον τρόπο εργασίας. Είχαμε επίσης ε, τους εκπροσώπους ελληνικής Task Force που μας εξήγησαν ότι στην Ελλάδα ήδη υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για αυτό το μέσο. Υπάρχουν έργα, προγράμματα που περιμένουν να τεθεί σε λειτουργία αυτό το μέσο. Συνεπώς είναι το θέμα πάρα πολύ κατεπήγον. Σχετικά με την ουσία συζητήσαμε ήδη το θέμα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Όπως ξέρετε είναι ένα μέσο κατά της κρίσης, ένα μέσο το οποίο θα διευκολύνει την ε, χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που αποτυγχάνει λόγω του γεγονότος ότι η ιδιωτική πόρη, η ιδιωτική χρηματοδότηση που χρειάζεται για ε, τέτοια έργα και προγράμματα ε, μαζί με την, τη δημόσια χρηματοδότηση δεν υπάρχει λόγω του κινδύνου, λόγω της έλλειψης διαθεσιμότητας τέτοιων ιδιωτικών πόρων. Γι' αυτό το μέσο αυτό το οποίο θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αυξήσει την ικανότητα να δίνει εγγυήσει και επίσης να παρέχει δάνεια, θα μπορούσε να διευκολυνθεί, να το μέσο αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει την κατάσταση για να έχουμε αυτά τα πρόσθετα κεφάλαια τα οποία λείπουν. Και αυτό κυρίως ε, για έργα υποδομών, αλλά επίσης ε, ε, στον τομέα του περιβάλλοντος, κυρίως στην Ελλάδα, Γι' αυτά ε, τα προγράμματα και έργα που προβλέπονται ήδη για αυτό το μέσο έχουν ε, σχέση με τα στερεά απόβλητα και θα, ο ρόλο, το μέσο αυτό θα ε, είναι ένας ε, ρόλος, θα έχει ένα ρόλο που θα διευκολύνει την πρόσβαση ε, στην ιδιωτική χρηματοδότηση. Θα υπάρξουν πολύ περισσότερα κεφάλαια για τα έργα που έχουν μπλοκαριστεί σήμερα. Το μέσο αυτό θα χρησιμοποιήσει τις δεσμεύσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 2007-2013 διότι υπάρχει ανάληψη, υπάρχει ανάληψη υποχρεώσεων, αλλά τα χρήματα δεν έχουν ξοδευτεί, δεν υπάρχουν πληρωμές από την πολιτική συνοχή. Έχουμε διευκρινίσει στην τεχνική συνεδρίαση και το Δεκέμβριο πάρα πολλά τεχνικά θέματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ε, θα έρθει σήμερα εδώ. Αν έχουμε και άλλες ερωτήσεις να τις θέσουμε. Από τη δική μου πλευρά, αυτά είναι τα βασικά ενημερωτικά θέματα. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι υπάρχουν δύο θέματα που είναι ανοιχτά. που είναι στην γνωμοδότηση που ετοιμάζει η ΕΚΟΝ η Επιτροπή Οίκων, συνάδελφο από την Επιτροπή Οίκων. Η πρόταση της Κομισιόν παρά τον τίτλο που είναι αρκετά ευρύσα στο κείμενο αναφέρεται στους τομείς της πολιτικής συνοχής στην χρηματοδότηση για τα έργα και προγράμματα τα οποία εντάσσονται στην πολιτική της συνοχής και αυτή η πρόταση όπως και η προηγούμενη Οκτωβρίου-Νοεμβρίου αναφέρεται στην συγχρηματοδότηση το ΠΑΠ με βάση τη νομική βάση, την κάλυψη γεωγραφική, τα προγράμματα βοήθειας που καλύπτουν έξι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι λοιπόν θα διευκολύνει το μέσο αυτό τους κανονισμούς για τις έξι χώρες ε, που χρησιμοποιούν το μέσο για το ισοζύγιο πληρωμών και που μπορούν να προσφύγουν στο EFSF οι 15 η Ευρωζώνη. Έχουμε ιδέες που ανακύπτουν. Γιατί να μην δημιουργηθεί με τα ευρωπαϊκά κονδύλια ένα μέσο το οποίο θα επέτρεπε τη χρήση για αυτού του είδους τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται μόνον εθνικά από δημόσιους πόρους και όχι από την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική και γιατί να μην επεκταθεί και σε άλλες χώρες που <clears throat> δεν εντάσσονται στα προγράμματα μακροοικονομικής βοήθειας, αλλά και σε άλλες χώρες που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο. Η Κομισιό είναι της γνώμης ότι δεν είναι καλή ιδέα, διότι οι δυνατότητες της Κομισιό να αντιμετωπίσουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αυτό το ευρύτερο σχήμα, ε, το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του μέσου, δεν της το επιτρέπει. Έχουμε βεβαίω πόρου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην πολιτική συνοχή. Αν επεκταθούμε λοιπόν ε, σε άλλου τομεί ε, επενδύσεων σε υποδομές, ε, τότε η πολιτική συνοχή δεν θα είναι η προτεραιότητα. Και χρησιμοποιώ τώρα τα επιχειρήματα τα οποία προέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε λοιπόν ε, στην Επιτροπή μας το έργο να λάβουμε απόφαση. Ίσως θα ζητήσουμε από την Επιτροπή και την Τράπεζα πρόσθετα επιχειρήματα, αλλά αυτά τα θέματα είναι ανοιχτά και τα αφήνω ε, στη δική σας συζήτηση. Θα πρέπει... Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την τρέχουσα κατάκταση, ε, την δυνατότητες της Κομισιόν, της υπάρχουσες, διότι αυτό ε, θα είναι ένα, ένα σχήμα, ένα μέσο το οποίο θα το διαχειρίζεται ε, κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Θα χρειάζεται λοιπόν προσωπικό από την DG, από την Γενική Διεύθυνση Ρίτζο και θα ήθελα εδώ να ζητήσω από, τους, από την κυρία Κλέβερ, την σοσιαλίστρια συνάδελφο, η οποία δραστηριοποιήθηκε για την προπαρασκευαστική εργασία. Θα ήθελα να τη ζητήσω τα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία και τη διοργάνωση της τεχνικής ενημέρωσης briefing εξαιρετική ενημέρωση αυτό το briefing. Τα περισσότερα ζητήματα αποσαφινίστηκαν και από πλευρά μου και από πλευρά των σοσιαλιστών θα είμαστε λοιπόν υπέρ της ταχύτερης επισπεσμένης διαδικασίας έγκρισης αυτού του εγγράφου από πλευρά μας. Το επόμενο σημείο για τη συνάντηση συνεδρίαση της οικων που συζητήθηκαν αυτά. Υπάρχουν πολλές παρερμηνίες ή θέματα που εκκρεμούν. Υπάρχει αυτή η έκθεση που δεν είμαι σίγουρη πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, διότι θα έχουμε και τη δική μας γνωμοδότηση. Θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. Ουσιαστικά για τις συζητήσεις εκεί θα μπορούσα να πω <clears throat> πρέπει να δούμε τι είναι επιλέξιμο και τι μπορεί να γίνει σε σχέση με αυτά τα εγχειρήματα, με αυτά τα σχέδια και για την πολιτική συνοχή, να μην επεκταθούμε σε όλα τα άλλα περαιτέρω. Συμφωνώ να επικεντρωθούμε σε αυτά. Είναι σαφές ότι τώρα αυτός ο μηχανισμός δεν είναι τίποτα το καινούριο. Είναι κάτι το γνωστό που όπως είπατε έχει ξεκινήσει. Ήταν μία από τις ανησυχίες που είχα. Δηλαδή αν θα ήταν κάτι καινούριο και δεν γνωρίζαμε το τι θα γινόταν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας επεξηγήσει τα πάντα τι περί τίνος πρόκειται, είναι, ποιοι είναι οι στόχοι και φυσικά ποιοι είναι οι, ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι στόχοι για την Ελλάδα. Να εγκριθεί λοιπόν το δυνατόν ταχύτερα, με το δυνατόν λιγότερες περιπλοκές είναι η άποψή μου. Είναι κατεπήγον. Να υποστηρίξουμε λοιπόν το, τους στόχους της Επιτροπής. Το επόμενο που θα ήθελα να πω είναι ότι κατά το μάλλον ήτον. Και θα ήθελα να ρωτήσουμε και τον Δανέζο, τον Δανό Υπουργό γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Συμβούλιο. Δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό, αν αυτό έχει κάποια πολιτική εξήγηση και ίσως δεν είναι κάποια προτεραιότητα. Ας το συζητήσουμε στο επόμενο σημείο, επίσης της ημερήσιας διάταξης με τον Δανό Υπουργό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, η κυρία Μανέσκου παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι προφανές ότι αλλάζοντας η αλλαγή του κανονισμού είναι σημαντική υπόθεση καθώς θα διευκολύνει την εφαρμογή των προγραμμάτων για τη συνοχή και θα έχει άμεση επίπτωση στις οικονομίες των κρατών μελών, ιδιαίτερα εκείνες τις οικονομίες που έχουν ιδιαίτερα πληγή από την κρίση. Έχω υπόψη την Ελλάδα ιδιαίτερα. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τη σημασία, τη σπουδαιότητα αυτού του επιμερισμού κινδύνου, αυτού του μέσου επιμερισμού κινδύνου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι το έγγραφο που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ τεχνικό χαρακτήρα, θα πρέπει να αναλύσουμε σε βάθος τους όρους, την ορολογία και τις προϋποθέσεις και όρους υπό τις οποίες και οποίους θα λειτουργήσει αυτό το μέσο, ώστε να είναι απόλυτα διαφανές, να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και να δούμε συγκεκριμένα χειροπιαστά δηλαδή πώς τέτοιου είδους μέσα θα επιτρέψουν να υπάρξει επιμερισμός ε, των κινδύνων. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, οι αρχές των κρατών μελών, το εκτελεστικό δηλαδή, θα χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια με το σωστό τρόπο. Συμφωνώ με την διαδικασία επίσπευσης, την ταχύτερη διαδικασία ή την κατεπίγουσα διαδικασία για να διευθετηθεί αυτό. Αλλά υπό τους όρους και προϋποθέσεις του να εξετάσουμε πολύ α, εκ του σύνεγγις ποιοι όροι θα εφαρμοστούν σε αυτόν τον επιμερισμό κινδύνων. Ευχαριστώ. Η κυρία Σρέτερ παρακαλώ. Καταρχήν συμφωνώ πρέπει να πω με την άποψη ότι είναι σκόπιμο αυτό το μέσο να το περιορίσουμε σε αυτό το πλαίσιο, ακριβώς όπως το έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το πεδίο. Δεύτερον, δεν είναι απόλυτα σαφές για μένα τι σημαίνει απλουστευμένη διαδικασία. Θα έλεγα το κείμενο όπως έχει υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανεπαρκές. Και επειδή είναι ανεπαρκές, γι' αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι αναγκαίο να καταθέσουμε τροπολογίες για να συμπληρωθεί εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε και οι πράσινοι θα καταθέσουν τροπολογίες από ό,τι γνωρίζω. Και αν αυτό μέσα στο πλαίσιο της επισπευμένης ταχύτερης διαδικασίας μπορεί να γίνει, τότε συμφωνούμε. Αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα. Και ζητώ και πάλι συγγνώμη που τώρα πρέπει να πάω σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή, που ήμουνα σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Σα συγχαίρω για την επανεκλογή σα ω πρόεδρο, κυρία Χούμπνερ, και την επανεκλογή των προέδρων. Σα ευχαριστώ εξ και όλων των αντιπροέδρων και εμού. Σα ευχαριστώ πολύ, Ελισάβετ. Ο κύριος Μπλάσκεκ έφυγε ήδη για άλλη επιτροπή. Α, εδώ είναι, εδώ είναι λέτε. Α, εκεί είσαστε, συγγνώμη, μετακινηθήκατε σε άλλο έδρανο. Εντάξει, έχετε τον λόγο λοιπόν. Já se omlouvám, došlo tady posunu k eh, přesazení, já nemám nějaký další komentář, abych chtěl využít. se ευχαριστώ. Αλλάξαμε θέση. Yeah, just... Θα ήθελα να συγχαρώ την, το νέο Προεδρείο. Σας εύχομαι ούριο άνομο και πάρα πολλές επιτυχίες στις διαπραγματεύσεις της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, είναι εδώ ο συνάδελφος. Χωρίς μικρόφωνο η παρέμβαση. Sorry, sorry. Can you Πρόεδρος, λοιπόν, αφού δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, αν δεν υπάρχουν... Α, εντάξει, εσείς κύριε Φανίστερ Ρόι, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ουσιαστικά είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων την τελευταία φορά στην Επιτροπή μας ήδη, δύο φορές ήδη. Και χαίρομαι που αναλώσατε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποσαφινιστούν όλα αυτά τα πράγματα και να επικαιροποιηθούν για ενημέρωση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε το δυνατόν να το κρατήσουμε αυτό μέσα στο πλαίσιο του κανονισμού, των κανονισμών για την πολιτική συνοχή και για την χρήση των κονδυλίων των ταμείων, των διαθροτικών ταμείων. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε συζήτηση που αφορά πάρα πολλά θέματα, έλεγχο προπολογισμού και άλλα. Άποψή μου λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να το κάνουμε και το υποστηρίζω. Σε ένα περιορισμένο πεδίο ή πλαίσιο για τα κονδύλια αυτά και τη διάθεσή τους και έτσι να απελευθερωθούν για αυτά, τα για τα σχέδια για το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες αν πρέπει αλλού να χρησιμοποιηθούν, όμως αυτό δεν μπορεί να μας απασχολήσει τώρα εδώ. Δεν είναι δική μας δουλειά για, τη, για τους κανονισμούς για την επόμενη περίοδο μπορούμε σίγουρα όλα αυτά να τα συζητήσουμε για να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία όσον αφορά τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των κονδυλίων. Εντάξει, η προσωπική μου άποψη είναι να σας υποστηρίξω όσον αφορά το ρόλο της εισηγήτριας που έχετε από την Επιτροπή μας για να γνωμοδοτήσετε και να μπορέσει το Συμβούλιο να προσελκυστεί και να ακολουθήσει τη δική μας στάση. Να μην αναμείνουμε για το Συμβούλιο ε, και το τι πρόκειται εκείνο να κάνει, εμείς να το επηρεάσουμε. Και για τη Δανέζικη Προεδρία είχαν πάρα πολλά κίνητρα, ιδιαίτερη κινητοποίηση για να το θέσουν αυτό ε, και με ε, επίσπευση να προχωρήσει και να λειτουργήσει. Αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη απόφαση. Ο κύριος Σταυρακάκης παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ξανά να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή σας και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Επιτροπή για την κατάθεση της πρότασης τροποποίησης που συζητάμε σήμερα. Μια πρόταση που έρχεται να δώσει μια απάντηση λύση στην επιδείνωση των προβλημάτων ρευστότητα και πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στι έξι χώρε που αναφέραμε. Μια πρόταση που χρησιμοποιεί τι υπάρχουσε δυνατότητε προκειμένου να καταστεί δυνατή υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομή που παραμένουν στάσιμα με τη χρηματοδότηση και την κινητοποίηση κεφαλαίων μέσω σχετικού μηχανισμού χορήγησης δανείων ή εγγύσεων. Όσον αφορά την κατάσταση στη χώρα μου, την οποία γνωρίζω πολύ καλά, η εφαρμογή των προτάσεων τη Επιτροπής θα βοηθήσει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση των έντονων προβλημάτων παροχής τραπεζική χρηματοδότηση λόγω τη κρίση και τη έλλειψη ρευστότητα. Πρακτικά έχει σταματήσει η υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων στη χώρα, τα οποία διαφορετικά θα μπορούσαν να δώσουν μια σημαντική αναπτυξιακή πνοή στην ελληνική οικονομία. Από τα πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και του σχετικούς υπολογισμούς οικονομολόγων προκύπτει ότι μέρος της σημερινής ύφης στην ελληνική οικονομία οφείλεται κατά 30% περίπου στην αδυναμία χρηματοδότησης των προγραμμάτων σχηματισμού παγίου κεφαλαίου σε υποδομές και άλλα αναπτυξιακά έργα. Ειδικότερα έργα που έχει προγραμματίσει ο δημόσιο τομέα δεν ξεκινούν ή έχουν σταματήσει καθώ η τραπεζική χρηματοδότηση δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί κάτω από τι τρέχουσε συνθήκε πιστοτική η πρόταση λοιπόν της επιτροπής έρχεται να δώσει λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα και προσφέρει την ευκαιρία επανεκκίνησης σημαντικών αναπτυξιακών έργων ενώ παράλληλα δεν έχει καμία επίπτωση στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. κλείνοντα θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ζωτική σημασία να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η πρόταση αυτής τη Επιτροπής. ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα τώρα να διακόψουμε λίγο τη συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε μετά τη συνεδρίαση, με την, την συνάντηση με τη Δανέζικη Προεδρία. Γιατί πρέπει να υπάρξει χώρο για του υπουργού να αποχωρήσουν οι βουλευτέ από εδώ, οι ευρωβουλευτέ. Διακόπτουμε συζήτηση για αυτό το σημείο. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα πλήρω και θα έχουμε και την Επιτροπή και άλλους συναδέφους που θα απαντήσουν. Θα παραμείνουμε στην αίθουσα, ε, προσέρχεται η Δανέζικη Προεδρία. Δεν αλλά για πρώτη φορά που στην άλλη αυτό που Τα το ξέρουμε αυτό. Αν κάτι λένε οι έχουν

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, επίσης προς τους βοηθούς και πολιτικούς συμβούλους και τα λοιπά και λοιπούς, ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας πάλι. Συνεχίζεται η συνεδρίαση, καθίστε παρακαλώ. Όπως γνωρίζετε, υπό αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης θα έχουμε τη συνάντηση με τον Υπουργό κύριο Νικολάη Βάμεν που εκπροσωπεί φυσικά την Δανέζικη Προεδρία του Συμβουλίου. Το χατοφυλάκιό του καλύπτει σχεδόν τα πάντα ως υπουργό που είναι Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Συντονίζει το έργο συνολικά της Προεδρίας Αρμοδιότητά του όμως είναι επίσης το πεδίο πολιτικής που αφορά την δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Γι' αυτό είναι σημαντική συνάντησή μας μαζί του σήμερα. Θα κάνουμε όπως συνηθίζουμε, θα ακούσουμε πρώτα δηλαδή τον Υπουργό και μετά θα έχουμε ερωτήσεις, σχόλια, αιτήματα που θα διατυπωθούν από τους Ευρωβουλευτές από εσάς. Έχουμε κάτι παραπάνω από μια ώρα για αυτή τη συνάντηση και ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρόνο αποτελεσματικά, με χρήσιμο τρόπο δηλαδή πραγματικά. Κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε. Έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Well, thank you. Μάλιστα, σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συγχαίροντά σα Πρόεδρε για την εκλογή σα ε, ω Πρόεδρο και πάλι στην Επιτροπή σα. και σα ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, τα καλά σα λόγια. Αγαπητοί συνάδελφοι, σα ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία να συναντηθούμε και να συζητήσουμε το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Πολιτική για την συνοχή. Χαίρομαι που είμαι ενώπιον σας στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρουσιάσω το πρόγραμμα της Δανέζικης Προεδρίας και για τις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις για την πολιτική συνοχή από πλευράς μου. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω πάλι με κάποια γενικά σχόλια όσον αφορά τη Δανέζικη Προεδρία. Προτού δώσω μια πιο εξειδικευμένη περιγραφή για τις φιλοδοξίες και τους στόχους μας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Μετά από την εισαγωγή μου, από ό,τι ακούω και το εκτιμώ αυτό, θα έχουμε χρόνο για ανταλλαγή απόψεων. Προσβλέπω σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας, κύριοι ευρώβουλευτέ. Στρέφομαι τώρα στις κυριότερες προτεραιότητε για την Δανέζικη Προεδρία του Συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά. Τέσσερις είναι αυτοί, αυτές οι προτεραιότητες ω άξονε. Ευθύνη, υπευθυνότητα από την Ευρώπη πρώτον, δυναμική Ευρώπη πράσινη Ευρώπη τρίτον και τέταρτον μια ασφαλή Ευρώπη. Αυτή είναι οι τέσσερι άξονε προτεραιοτήτων. Σε σχέση με την πρώτη προτεραιότητα, υπεύθυνη, υπευθυνότητα από την Ευρώπη, είναι σαφές ότι πρέπει να αποκατασταθεί η τάξη και η σταθερότητα στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Παρότι η Δανία είναι εκτό Ευρωζώνη, εργαζόμαστε σκληρά για αυτή την ημερήσια διάταξη, για αυτά τα θέματα, όπου περνάει από το χέρι μα και όπου μπορούμε, στο ΕΚΟΦΗΝ και στα Συμβούλια για την ημερήσια διάταξη για την ανάπτυξη. Ουσιαστικά, συνάδελφοι, πρέπει να υπάρξει το δυναμικό ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να είμαστε γέφυρα μεταξύ Ευρωζώνη, κρατών μελών και μελών, κρατών μελών εκτό Ευρωζώνη σίγουρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαντήσει αποτελεσματικά και με πιστικό τρόπο, με πειθό, ώστε οι άμεσες απειλές ε, λόγω του ανέφικτου, του αδύνατου να αντιμετωπιστεί χρέους σε κάποιες οικονομίες, να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτό, απαιτεί βούληση και συμμόρφωση με νέους κανόνες για την οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση και διαχείριση που αποτελούν τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτοί οι κανονισμοί και κανόνες θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της Δανέζικης Προεδρίας. Μια άλλη προτεραιότητα θα είναι να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων όσον αφορά τον δημοσιονομικό, τους δημοσιονομικούς κανονισμούς και Αυτό είναι αναγκαίο για ένα ε, υγιές ε, τραπεζικό σύστημα και για την ελαχιστοποίηση μελλοντικών κρίσεων. Το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα βρίσκεται πάνω-πάνω στην ημερησία διάταξή μα. Είναι ζωτική σημασία να διαθέσουμε με ένα προπολογισμό νέα κονδύλια, αυξημένα κονδύλια για την έρευνα, ανάπτυξη και την πράσινη, πράσινες τεχνολογίες. Κατά του πρώτου μήνε τη προεδρία μα, ελπίζουμε ότι θα αποσαφηνίσουμε πολλέ τεχνικέ πτυχέ επ' Δεύτερον, καθώ θα συνεχίζουμε, θα κινηθούμε σε μια πιο πολιτικού χαρακτήρα φάση, όπου θέλουμε να μειώσουμε το χάσμα και τη διαφορά μεταξύ των διαφορετικών τοποθετήσεων και θέσεων των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινή μαζί σα. Δεν είναι ρεαλιστικό να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει, να πιστεύει κανεί ότι θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει υπό την Δανέζικη Προεδρία. Ελπίζουμε όμω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλέ θέσει και προτάσει για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει, το δυνατόν περισσότερα θέματα να ολοκληρωθούν πριν από το τέλο ε, τη δική μα Προεδρία. Γίνονται προσπάθειες για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα δημοσιονομικά από τις κυβερνήσεις, τα κράτη-μέλη. Πρέπει να δούμε, να έρθουμε στο ύψος των ευθυνών και ευ, της ευθύνη μας και πρέπει έτσι να διαμορφωθεί η μερίσια διάταξη. Όμως για τον πολιετή προϋπολογισμό για την Ευρώπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μόνο θέμα περικοπής δαπανών, περιστολής δαπανών. Πρέπει να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Αυτή η φιλοδοξία πρέπει να αντανακλάται απόλυτα και πλήρως στον προϋπολογισμό μας δημοσιονομικά. Οι δημοσιονομικές αυτές ευθύνες για την ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης πρέπει να βαίνουν εκ παραλίλου. Δεύτερη προτεραιότητα, να επανέλθει η Ευρώπη σε έναν μια πορεία ανάπτυξης. Αυτό συναρτάται με την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Εφέτος θα έχουμε την 20η επέτειο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς αποδείχθηκε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα ιστορικά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο δυναμικό που παραμένει ανεκμετάλλευτο ακόμα και στόχος της, Ευρωπαϊ... της Δανέζικης Προεδρίας είναι να συνεισφέρουμε να εκπληρωθεί, να αναπτυχθεί και να εξυγχρονιστεί αυτό το δυναμικό, αυτή η δυνατότητα, βελτιώνοντας το κλίμα ε, το επι... του της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, εξυγχρονίζοντας και επικαιροποιώντα ε, τους κανονισμούς για τις επιχειρήσεις ε, για τα κεφάλαια κινδύνου, καθώς και πιο ευέλικτους κανονισμούς και κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες. Επίσης, θα έχουμε καλύτερη, μεγαλύτερη ασφάλεια online διαδικτυακά για τους ε, καταναλωτές όταν ε, αυτοί κινούνται διαδικτυακά και μέσω επικοινωνιών. Θέλουμε να προσαρμοστεί μια πιο φιλόδοξη, ε, ένα πιο φιλόδοξο εγχείρημα για το πρασίνισμα της οικονομίας. Καθώς εμπλεκόμαστε στη διαχείριση της κρίσης, η ευρωπαϊκή οικονομία, οι ευρωπαϊκές οικονομίες πρέπει να είναι αηφόρες μακροπρόθεσμα έχει πρωτοπόρο ρόλο η Ευρώπη παγκόσμια στην πράσινη ατζέντα, αναπτύσσοντας μια ε, σχετική πρωτοβουλία και για το πρασίνισμα. Τώρα πρέπει να επιταχύνουμε το πέρασμα στην Ευρώπη σε μια πράσινη και πιο αηφόρα οικονομία. Ο τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε είναι δημιουργώντας θέσεις, ε, ε, απασχόλησης και ανάπτυξης, χωρίς να ε, ακολουθήσουμε πορεία εκμετάλλευση ορυκτών καυσίμων, να εγγράψουμε θέματα στην ημερήσια διάταξη με μεταρρύθμιση και μεταρρυθμίσει ε, για την ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική, αλλιευτική πολιτική, Πρέπει όμως να είμαστε και ρεαλιστές από την άλλη πλευρά. Έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα, δεν θα τα καταφέρουμε αυτόματα όλα αυτά και από μόνα τους. Πρέπει να συνεργαστούμε για τις πράσινες πρωτοβουλίες αν θέλουμε να διατηρήσουμε τα συγκριτικά προτερήματά μας σε σχέση με άλλες περιφέρειες και υπήρους παγκόσμια. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο ε, θέσεις απασχόλησης λόγω της μετακίνησης της γνώσης και της τεχνογνωσίας να μετατεθούν σε άλλες υπήρους ε, σε σχέση με την μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία. Η πράσινη μεταφορά και μετάθεση πολλά σημαίνει, αλλά το να προλιάνουμε το έδαφος μακροπρόθεσμα για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη είναι ένα τμήμα αυτής της προσπάθειας. Δεν είναι μόνο το να δημιουργηθούν κάποιοι ευνοϊκοί στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε μετά από 30 χρόνια. Θέλουμε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης που θα βασίζονται στη γνώση βραχυπρόθεσμα στην Ευρώπη. Η Δανέζικη Προεδρία θα δουλέψει σκληρά για την προαγωγή αυτής της πράσινης ατζέντας ημερήσιας διάταξης. Αλλά θα πρέπει να είναι με έναν τρόπο συνολικό συνολικό που θα γίνει αυτό που θα κινητοποιήσει τους πάντες. Τέταρτη προτεραιότητα, πιο ασφαλής Ευρώπη. Θα θυμόσαστε, οι πρώτοι μήνες ε, της ε, Αραβικής Άνοιξης ανάγκασαν χιλιάδες Αφρικανούς να μετακινηθούν στην Ευρώπη αναζητώντας ε, καταφύγιο και προστασία. Αυτά τα προβλήματα με την παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη υπογραμμίζουν την ανάγκη να ολοκληρώσουμε μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για μια κοινή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο, ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται σωστά αυτοί που προσέρχονται στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο. Μια λειτουργική πολιτική για το άσυλο, μια πιο ενισχυμένη πολιτική συνεργασία μέσα στα πλαίσια του Σέγγεν. Λοιπόν, η πολιτική συνοχή, πού ταιριάζει μέσα σε αυτό το πλαίσιο για τη Δανέζικη Προεδρία. Επιτρέψτε μου παρακαλώ να σας υπενθυμάσω, να σας υπενθυμίσω με συγχωρείτε τις ιστορικές ε, πρόπτικες. Το 2002 το φθινόπωρο είχαμε την ε, Προεδρία Δανία όταν αποφασίστηκε η διεύρυνση. Η πολιτική συνοχή είχε, έχει και συνεχίζει να έχει, θα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης της σύγκλησης και συνοχής σε σχέση με την Ήπειρό μας που αποφασίστηκε να επανενωθεί πλέον μέσα σε αυτό το πλαίσιο στην Κοπενχάγη το 2002. Διανύσαμε μεγάλη πορεία, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο ακόμη. Όπως ήδη προανέφερα στην εισαγωγή μου, αντιμετωπίζουμε οικονομικές συνθήκες που θα εξακολουθήσουν να είναι πάρα πολύ προκλητικές, μεγάλες προκλήσεις. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε όπως στο παρελθόν, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα. Όμως σε σχέση με αυτή τη θέση συνένεσης Ευρώπης και η δημοσιονομική πίεση μας αναγκάζει να κινηθούμε προς μια ενιαία κοινή πορεία. Πρέπει να συνεργαστούμε για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη, η αύξηση, η οικονομική αύξηση της Ευρώπης, ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Σε σχέση με την οικονομική κρίση θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής είναι μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας και επιτευγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο σύμβολο ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά επίσης αντανακλά θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και ταυτόχρονα είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο να προπαρασκευαστεί η Ευρώπη για τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτά τα σκεπτικά, αυτές οι σκέψεις είναι τα θεμέλια και η βάση της Δανέζικης Προεδρίας στον τομέα της πολιτικής συνοχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως εσείς περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλους έχετε συνειδητοποιήσει, η πολιτική συνοχή σήμερα είναι αντικείμενο κανονικής νομοθετικής διαδικασίας και εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν κοινέ ευθύνε από κοινού ω συνομοθέτε να προαγάγουν την πολιτική συνοχή μέχρι το 2020. Και αυτό είναι ένα έργο στο οποίο πρέπει να συνεργαστούμε όλοι από κοινού. Και η Δανέζικη Προεδρία καλωσορίζει την ευκαιρία να συνεργαστεί εκ του σύνεγγυ πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα, ομιλώντας για το 2020, κύριε και κύριοι, Επιτρέψτε μου παρακαλώ να υπενθυμίσω ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεών μας με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν τη στρατηγική για τους στόχους για την Ευρώπη του 2020. Αηφορία, ανάπτυξη συνολική, και σε σχέση με τα συμπεράσματα του Μαρτίου 2010 είπε το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο ότι οι προσπάθειές μας πρέπει να επικεντρώνονται με καλύτερο τρόπο σε πιο συντονισμένη στοχοθέτηση για αυξημένη ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, δυναμικό για την ανάπτυξη και οικονομική σύγκληση και συνοχή. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επίσης συνεπέραναν ότι όλε οι κοινέ πολιτικέ, συμπεριλαμβανομένε και τη πολιτική συνοχή, θα πρέπει να υποστηρίζουν του στόχου επίτευξη τη στρατηγική του 2020. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο δρούμε και λειτουργούμε. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό και σε σχέση με τι αποφάσει που θα πρέπει να ληφθούν δημοσιονομικά. Οι που έχουμε έχουμε ενώπιόν μα είναι λοιπόν να βρούμε, να εξεύρουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα επικεντρώνεται με αυτόν τον τρόπο στου στόχου που εξέθεσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Όμω επαρκώ προσαρμόσιμο στις συνθήκε και προποθέσει επιτόπου, στο πεδίο. Ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να υπεκφύγουμε, να απεμπολίσουμε τι ευθύνε του να αρθούμε στο ύψο των περιστάσεων να απαντήσουμε στα εξή ερωτήματα. Πώς μπορούμε από κοινού να συνεισφέρουμε με ένα στοχοθετημένο τρόπο στην αντιμετώπιση αυτών των στόχων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δώσουμε αξία για τα κονδύλια και τα χρήματα που δαπανούμε. Η πολιτική συνοχή πρέπει να είναι στοχοθετημένη και με σωστού προσανατολισμού. Το ίδιο ισχύει και για την διαδικασία διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων. Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ανάγκη να καταδείξουμε ότι λειτουργεί, λειτουργεί σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η κοινοτική μέθοδο λειτουργεί και λειτουργεί σωστά και ότι είμαστε σε θέση να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα προ όφελο των πολιτών μα. Για μας, για λογαριασμό μα θέλουμε να προαγάγουμε τι διαπραγματεύσει στο μέτρο του εφικτού. Και μέσα αυτά τα πλαίσια ας είμαστε ειλικρινεί και ομοί. Με ομότητα και ειλικρίνεια να το πούμε αυτό και να το πούμε εξάπαντος. Οι καθαροί πληρωτές ε, όπως ε, η Δανία σε σχέση με κάποια επιχειρήματα για την μη προαγωγή της πολιτικής συνοχής ότι δεν θα υπήρχε λέει ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Λάθος αυτό. Το αντίθετο συμβαίνει ακριβώς το πακέτο, το δέσμη μέτρων για, τα, για τη συνοχή είναι τόσο σύνθετο και περίπλοκο που δεν μπορούμε να αναμείνουμε να δούμε τι γίνεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να δούμε τι γίνεται με άλλους. Προτού ξεκινήσουμε τη δράση μας. Προφανώς αυτό και πάλι είναι προς όφελος και θα είναι προς όφελος των αποδεκτών των πολιτών επιτόπου στο πεδίο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, θα πιέσουμε να σημειωθεί πρόοδος. Αποκινούμε όλους εσάς να προχωρήσουμε, να επιτευχθεί πρόοδος, να σημειωθούν χειροπιαστές στα αποτελέσματα. Η Δανέζικη Προεδρία στοχεύει στο να προβεί σε μια εκπαραλλήλου ανάπτυξη και πορεία προς αυτή την επίτευξη αυτών των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν στο τέλος. Προφανώς η νομοθεσία για την πολιτική συνοχής δεν μπορεί να ολοκληρωθεί παρά μόνο μέχρι ότου εξευρεθεί τελική συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Σε σχέση με την πορεία για το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, το Συμβούλιο το Δεκέμβριο ήταν σαφέστατο όταν ζήτησε από την επόμενη Προεδρία να συνεχίσει τις προσπάθειες ε, με βάση το έργο που είχε επιτελεστεί για να ολοκληρωθούν οι τελικές φάσεις διαπραγματεύσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο 2012. Και όλα αυτά τι συνεπάγονται. Συνεπάγονται ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής όλοι μας όλοι μας έχουμε κάθε συμφέρον να παραμείνουμε σε αυτή την πορεία και να συνεχίσουμε και να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε, να προσαρμοστούμε σε νέα στοχοθέτηση και τις προκλήσεις και να πετύχουμε. Η Δανέζικη Προεδρία συνεχίζει στα καλά θεμέλια που έθεσε η Πολωνική Προεδρία. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε στις διαπραγματεύσεις να σημειωθεί πρόοδος. Λάβαμε πραγματικά μια ε, υποστήριξη και μια νέα όθηση που δόθηκε σε σχέση με το Συμβούλιο και σε σχέση με το Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων τον Ιούνιο θέλουμε να έχουμε προχωρήσει. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας όμως. Χρειαζόμαστε το Ευρωκοινοβούλιο ως στενό μας ε, εταίρο, στο πλευρό μας, για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στη σωστή πορεία σε αυτό το σύρμο, το τρένο που ακολουθεί αυτή τη διαδρομή. Όχι μόνο να ακολουθήσουμε τη σωστή πορεία, αλλά τα διαφο οι διάφοροι σειρμοί να μην ακολουθήσουν διαφορετική τροχιά, να μην ακολουθηθεί διαφορετική πορεία παρεκκλίνοντα από οποιονδήποτε. Πρέπει τώρα να συνεχίσουμε την πορεία. Είμαστε συνομοθέτε. Έχει σημαντική επιρροή αυτό στον βαθμό που μπορεί να επιτευχθεί πρόοδο ε, προ όφελο και προ το συμφέρον των χωρών μα. Η δανέζικη κυβέρνηση λοιπόν έδωσε εντολή στου εκπροσώπου τη Δανία εδώ στι Βρυξέλλε να βρίσκονται σε πολύ στενή ε, συνεργασία συνεργασία και επαφή με το Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να είναι ε, δυνατόν να υπάρχει ενημέρωση, να συζητώνται τα θέματα σε διαβούλευση και να υπάρχει απόλυτη ενημέρωση, ώστε να αποφευθεί παρέκκληση μεταξύ των συνομοθετών και να βελτιωθούν οι πιθανότητε και οι ευκαιρίες να επιτευχθεί συμφωνία το δυνατόν ταχύτερα. Κυρίε και κύριοι, ευελπιστώ ότι από κοινού μπορούμε να επιτύχουμε στις προσπάθειές μας αυτές από κοινού. Θα ήθελα μόνο κάποια σχόλια να κάνω σε σχέση με την ε, έγκριση του πακέτου των, της δέσμης μέτρων για, το, για τη συνοχή. Οι πρώτες εντυπώσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές. Αυτό συμβαίνει τόσο περισσότερο μια και αντιμετωπίζουμε με ένα, ένα ιδιαίτερα περίπλοκο και σύνθετο τμήμα νομοθεσίας. Πρώτον είναι πολύ εύκολο κανείς ε, να έχει κάποιες αρνητικές εντυπώσεις ε, και να μην προσαρμοστεί ή να μην καθορίζεται από την πραγματικότητα σε αυτά. Αυτό έχει σχέση με την ανθρώπινη φύση όσον αφορά τις αλλαγές που απαιτούνται. Οι αλλαγές οποίες όμως καμιά φορά είναι υποχρεωτικές για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις εξελίξεις. Αυτό είναι τόσο περισσότερο αναγκαίο σε αυτό το σταυροδρόμι που, στο οποίο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην μας τρομάζουν λοιπόν και μας ξενίζουν κάποιες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με τους όρους εξ άντε, εκ προημίου προϋποθέσεων, υλοποίησης ε, προϋποθέσεων και σε σχέση και με τη στρατηγική προσέγγιση στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού για την επίτευξη στόχων. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα συζητήσουμε συζητήσουμε όλα αυτά τους επόμενους μήνες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Υπάρχει εδώ και ένα μήνυμα για τις ε, προτινόμενες αλλαγές σε σχέση με την Επιτροπή και είμαι βέβαιος ότι θα εξεύρουμε πρακτικές λύσεις και θα επικεντρωθούμε στις σωστές λύσεις σε αυτό το οποίο φαίνεται ένα περίπλοκο και αξεδιάλειτο πακέτο μέτρων. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι τα υπόλοιπα είναι η, η ολοκλήρωση των λεπτομεριών ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε. Είμαι πεισμένο ότι είμαστε κάτι παραπάνω από ικανοί να τα πετύχουμε αυτά. Το μήνυμα που θέλω να σας δώσω σήμερα είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Και με το πνεύμα του ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όχι μόνο λέω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει βεβαιότητα. Από πλευρά του Συμβουλίου έχουμε αντιμετωπίσει τα θέματα τη απλούστευση, αντιμετωπίζουμε τα θέματα απλούστευση, διαχείριση μεγαλύτερων προγραμμάτων και σχεδίων και διαχείρισή του. Αξιολόγηση επίση των ε, επιτευγμάτων. Ακολουθούμε και συνεχίζουμε στα ισχυρά θεμέλια που ετέθησαν από την Πολωνική Προεδρία στον προγραμματισμό, σχεδιασμό και συντονισμό με συντονιστική συνεδρίαση που έγινε και χθε. Λοιπόν, στη σωστή χρονική συγκυρία θα πρέπει κάποια οριζόντια στοιχεία να τα λάβουμε υπόψη σε σχέση με την πολιτική του σημασία στο τέλος τέλος. Όπως είπα, η πολιτική συνοχή θα εγγραφεί σε δύο από τις συνεδριάσεις ε, του, του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου και τέλη Ιουνίου. Ε, με αυτές τις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής στην Ευρώπη θέλουμε να ολοκληρωθούν και οι διαπραγματεύσεις για οποιασδήποτε αλλαγές σε σχέση με το σημερινό πλαίσιο συνοχής. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εισαγωγή μέσων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Προτάθηκαν ήδη πέρυσι, το 2011. Κάποια κράτη-μέλη ήταν υπέρ του να δημιουργηθούν αυτά τα μέσα μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για να καταπολεμηθεί η κρίση πιο αποτελεσματικά με κάποια τύχη που χρειάζεται και απαιτείται και με επικοδομητικό πνεύμα συνεργασία θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε με αυτέ τι διαπραγματεύσει. Λίγο χρόνο απομένει. Πρέπει να είμαστε σοφοί και συνετοί στη χρήση του χρόνου για να είμαστε αποτελεσματικοί και να λάβει την καλύτερη διαμόρφωση, να διαμορφωθούν όλα αυτά στο καλύτερο πλαίσιο. Θέλω να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία για το εξαιρετικό έργο που επετέλεσε. Αυτό το κάνει, αν όχι εύκολο, επειδή δεν είναι εύκολο βέβαια το να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει, μια και έχουν τεράστια εμβέλεια, τουλάχιστον είναι πιο εύκολο να δούμε το φω στην άκρη τη στο τέλο τη σύραγγα. Και καθώ γνωρίζετε είχαμε μια ε, συνάντηση των Υπουργών Γενικών ε, Υποθέσεων που είχε ε, συγκληθεί τον Δεκέμβριο. Δεν μπορώ να πω ότι θα έχουμε την ίδια επιτυχία ως Δανέζικη Προεδρία. Μας βοήθησε όμως η πολωνική αυτή εκδήλωση να προχωρήσουμε και από αυτών των θεμελίων θα οικοδομήσουμε. Φαίνεται πιθανότερο ότι το κοινό στρατηγικό πλαίσιο στο τέλο τέλος θα προσαρμοστεί και θα επικαιροποιηθεί σε σχέση με την καθημερινή νομοθετική διαδικασία και ευελπιστώ ότι θα υπάρξει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού. Δεύτερον, ήταν επίσης απόλυτα σαφές ότι χρειαζόμαστε μια πολύ προσεκτικά προσαρμοσμένη προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο οι, ε, οι εξειδικευμένοι προσανατολισμοί ανά χώρα θα εφαρμόζονται για την πολιτική συνοχή. Δεν μπορούμε αφενός να διαχωρίσουμε την πολιτική συνοχή από τη συνολική πολιτική για τα οικονομικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, οι συστάσει δεν είναι πάντα αρκετά εξειδικευμένε για μια πολιτική επενδύσεων. Πολλέ φορέ αφορούν ε, μεταρρυθμίσει. Έχουν συστάσει που απευθύνονται στα κράτη-μέλη. Ενώ η πολιτική συνοχή βασίζεται σε κανονισμού και σε επιμερισμένη διαχείριση και τα περισσότερα διεξάγονται στο περιφερειακό επίπεδο και όχι σε κεντρικό επίπεδο. Αυτό διαφοροποιεί τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να εξεύρουμε αποδεκτέ λύσει για όλα αυτά τα θέματα. Μία συζήτηση για σημασιολογικά θέματα για τη σημαντική επικέντρωση και πιο ενισχυμένη επικέντρωση των κονδυλίων για την πολιτική συνοχή θα δώσει την δυνατότητα να αναθεωρηθεί η κριτική μάζα και να προσαρμοστούμε στι πολιτικέ επιτόπου, στο πεδίο. Ταυτόχρονα πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, απέχουν πόρο από το να έχουν συμφωνήσει επί όλων των λεπτομεριών. Δεν είναι ακόμα τα κράτη-μέλη να πούν ποια είναι η τελική του ε, ε, κόκκινη γραμμή και τι τελικά είναι πρόθυμοι να κάνουν ή όχι. Θα δούμε λοιπόν πώς αυτοί οι περιορισμοί, αυτές ε, οι ανάγκες θα καθορίσουν το έργο και τι θα, ποια θα είναι η τελική έκβαση. Η Δανέζικη Προεδρία θέλει να δώσει λίγο περισσότερο χρόνο για να οριμάσουν όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν τεράστια πολιτική σημασία και πολιτικό χαρακτήρα. Στο τέλος τέλος θέλουμε να οριμάσουν για να ευδοκιμήσουν. Στο μεσοδιάστημα κυρίες και κύριοι, στοχεύουμε να επιτελέσουμε πραγματική πρόοδο και να μπορέσουμε σε αυτούς τους ακρογωνιαίους λίθους ε, να θεμελιώσουμε το έργο μας. Απαιτείται πειθαρχία και ένα χρονοπλαίσιο στο οποίο θα ανταποκριθούμε. Ο χρόνο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Είμαστε όμω στα χέρια των αντιπροσωπιών όταν διοργανώνουμε και προσπαθούμε να διοργανώσουμε αποτελεσματικά τι διαπραγματεύσει μα. Στο τέλο τέλος η ε, πρόοδο εξαρτάται από την προθυμία όλων να ανταποκριθούν στι προκλήσει. Ανταπόκριση στι προκλήσει. Να είσαστε βέβαιοι λοιπόν ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα Να προαχθούν αυτέ οι διαπραγματεύσει στο μέτρο του εφικτού όσο γίνεται πιο σε αυτό το εγχείρημα προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία του σύνεγγυς με το Ευρωκοινοβούλιο. Πραγματικά πιστεύω στεναρά ότι από κοινού, ενωμένοι, με βούληση, με σθένος, με σκληρή δουλειά θα, τα καταφέρουμε και θα προχωρήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο προσβλέπει με συνεργασία σε εσά να επιτύχει η Δανέζικη Προεδρία στην πολιτική συνοχή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και σας ευχαριστώ που παρουσιάσατε την πολιτική συνοχή ως προτεραιότητα ε, για την Προεδρία σας ε, με αυτό τις προκλήσεις ε, και τα προβλήματα που έχουμε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και έτσι μπορούμε να δούμε καλύτερα τις σχέσεις με την υπόλοιπη δουλειά και το υπόλοιπο έργο το οποίο έχει να επιτελέσει η Ευρώπη. Ανοίγω την συζήτηση. Αρχίζουμε με τους συντονιστές για το El Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον Υπουργό για την παρουσίασή του που ήταν σαφής. Βεβαίως είμαστε φίλοι, αλλά μπορεί κανείς και να χάσει φίλους και λέει κανείς ότι ο χρόνος είναι φίλος μας, αλλά μπορούμε να χάσουμε και το χρόνο. Αυτή είναι μια έκφραση που έχουμε. Μπορεί να χάσουμε την προθεσμία του 2014. Αν χάσουμε αυτή την όθηση που μας οθεί προς μια πιο ολοκληρωμένη μέθοδο, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της στρατηγικής 2020. Αν πάμε προς τα πίσω, βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να στοιχηματίσουμε στο χρόνο. Ε, το βλέπουμε με τα όσα συμβαίνουν, ε, συνέβησαν στην Επιτροπή μας. Αναφέρατε αυτό το ρυθμό με τα διάφορα building blocks, αλλά βεβαίως ε, τα διάφορα δομοστοιχεία τα οποία πρέπει να μπουν στη θέση τους και αναφέρατε τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις διότι θα συνεχίσουμε με αυτές τις δυσκολίες και χάνουμε χρόνο. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών η Επιτροπή μας θα πρέπει να αναλύσει σαφώς αυτά τα διάφορα building blocks και στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να προβλέψουμε αυτούς τους κανονισμούς. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε και να προχωρήσουμε. Αυτό που με εκπλήσει είναι ότι διαπιστώνω ότι ε, δεν επαναλάβατε το ρυθμό της Πολωνικής Προεδρίας, δεν τον συνεχίζετε αυτό το ρυθμό. Ένας υπουργός επιφορτισμένος με την συνοχή δεν το έχετε αυτό στο πρόγραμμά σας. Δεν ξέρω αν προβλέπονται διασκέψεις, ε, σύνοδοι κορυφής, ε, επίσημοι ή ανεπίσημες, άτυπες ε, ίσως δεν παρακολούθησα πολύ καλά τα όσα είπατε, μήπως μπορείτε ακόμη να μας πείσετε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε, είμαστε υπεύθυνοι, υπεύθυνοι για ορισμένους φακέλους και θα πρέπει να συνεργαστούμε. Συνεπώς, Όλες αυτές οι ιδέες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά χτες στην Επιτροπή Ήτρε ο συναδελφός σας μας είπε ότι θα οργανώσει σεμινάρια, ε, διασκέψεις, συνέδρια για πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Ο κύριος Χάν ε, είναι ενδιαφερόμενος, έχουμε τα κέντρα αριστείας. Ε, για να υλοποιηθεί αυτή η ατζέντα του ορίζοντα 2020. Τι γίνεται με την ολοκληρωμένη προσέγγιση, μπορείτε να μας πείτε πώς εσείς ε, θα μας κάνετε να συμμετάσχουμε, έχουμε ένα ρόλο και πώς αντιλαμβάνεστε τη συνεργασία μαζί μας και τον προγραμματισμό μας. Χαιρόμαστε που αναφέρατε ενδείξεις ε, θετικές αυτό το στρατηγικό πλαίσιο, το κοινό πλαίσιο Έχουμε εδώ αρκετά να κάνουμε και πιστεύω ότι είναι χρήσιμο εσείς να είστε στο πλευρό μας και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε επίσης στα πλαίσια της παρέμβασης του κυρίου Χαν αφετέρου. Μου φαίνεται κάπως επιφυλακτικός σε σχέση με άλλες δυνατότητες. Μας λέτε ότι με λίγη τύχη ή με πολύ τύχη θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα νέα μέσα για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια της συνοχής μου φαίνεται ότι είναι ουσιαστικό να περιοριστούμε σε αυτό περί του οποίου πρόκειται στα θέματα αυτά καθεαυτά, να μην κάνουμε πιο περίπλοκο ένα φάκελο και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να γίνουν οι τελευταίες προσαρμογές αυτού του κανονισμού για να προχωρήσουν τα πράγματα. Αυτό βεβαίως απαιτεί πολλή τύχη, όχι μόνο λίγη τύχη. Αυτά. Αυτά. Αυτές είναι οι διάφορες παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω, γενικές παρατηρήσεις, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε με πιο συγκεκριμένα πράγματα. Θα ήθελα να ζητήσω από την Κωνσταντσα Κρίλεξ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε. Το χαιρετίζω ότι έχετε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσατε για την πολιτική συνοχή. Αλλά και αυτό είναι αναγκαίο. Αν θέλουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας σε πολλά πράγματα να μην σταματήσουμε και θέλουμε να επιτευχθεί πρόοδος, ε, πρέπει να επιταχύνουμε, να κινηθούμε προς τα εμπρός, γιατί αλλιώς το 2014 δεν θα τα καταφέρουμε. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε, ότι χρειάζεται αποτέλεσμα χειροπιαστό σε σχέση με τους προσανατολισμούς στην Προεδρία Κάποια σημεία θα ήθελα να αναφέρω από στις πρώτε συζητήσει που είχαμε εδώ στην Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή, όπου υπάρχει μια κατεύθυνση, ένα προσανατολισμό και όπου υπάρχουν και πλειοψηφίες για την τροποποίηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως έχει κατατεθεί, έχουμε αφενός το θέμα το ότι φυσικά υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εγχείρημά τη η πολιτική συνοχή να οδηγήσει στην επίτευξη και υποστήριξη των στόχων τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Απόλυτα σαφέ αυτό. Όμω η πολιτική τη συνοχή είναι κάτι πολύ παραπέρα και παραπάνω από αυτό και για τις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό αυτό δεν πρέπει να αμελείται, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ελπίζω ότι η Προεδρία σας και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και θα αναζητήσει χειροπιαστά αποτελέσματα στο τέλος τέλος. Αυτό τι σημαίνει για μας. Σημαίνει ότι σε κάποια σημεία πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ελαστικότητα από αυτή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά της μεγαλύτερη ελαστικότητα. Ξεκινήσαμε να συζητούμε αυτά τα θέματα στην κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Πιστεύω όμως ότι μια πλειοψηφία στην Επιτροπή μας είναι της άποψης ότι πρέπει να διοργανωθεί η δυνατότητα αυτής της ελαστικής δράσης, ελαστικής ε, ευέλικτης αντιμετώπισης. Και ένα πιθανό μέσο θα ήταν οι συμβάσεις και συμφωνίες εταιρικής σχέσης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που όμως στα σχέδια κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επεξηγεί επαρκώς και διεξοδικά ποιο καθεστώς θα έχουν και θα έχει και η ίδια Ξέρω ότι η συζήτηση στο Συμβούλιο εκ παραλίλου αναπτύσσεται όπως και αυτό. Θα θέλαμε όμως εμεί ως Ευρωκοινοβούλιο αυτέ οι συμβάσει και συμφωνίε εταιρική σχέση να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, ώστε στα κράτη-μέλη και στι περιφέρειές του να δίνεται η δυνατότητα να εμπλέκονται περισσότερο εκπροσωπώντα τα συμφέροντά του και έτσι να συνάπτονται αυτέ οι συμφωνίε και συμβάσει. Για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο αναφέρθηκαν αρκετά πράγματα, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εγώ εδώ. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω για άλλη μια φορά όμως είναι ότι οι διαπραγματεύσεις για την πολιτική συνοχή βαίνουν εκ παραλλήλου. πρέπει να βαίνουν εκ παραλίλου όπως και οι διαπραγματεύσεις για τη γεωργία και την αλληλεία, την κοινή αλληλευτική πολιτική και με τις διαπραγματεύσεις για την έρευνα που έχουμε. Διότι προσέχοντας όλα αυτά να ενταχθούν σε ένα κοινό σύστημα, θα πρέπει να μην κατακαιρματιστούμε και παρεκκλίνουμε στις διαπραγματεύσεις ανάλογα με το αντικείμενο όλα αυτά συνολικά να βρίσκονται σε ένα ενιαίο κοινό πλαίσιο και να λειτουργούν σωστά. Στο θέμα της απλούστευσης. Για την απλούστευση σήμερα το απόγευμα σίγουρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσουμε να συζητήσουμε σε βάθος περισσότερο για αυτά τα θέματα. Πρέπει να μεριμνήσουμε όμω και στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι μόνο στην επιφάνεια να παραμείνουμε και να υπάρχουν απλουστεύσει στο σύστημα διαχείριση, αυτέ οι απλουστεύσει να πάνε σε βάθο και να φτάνουν σε εκείνου που συντάσσουν τι αιτήσει για να του δοθούν κονδύλια και να υποστηριχθούν. Σε αυτούς πρέπει να φτάνουν τα αποτελέσματα. Δεν είναι το αποτέλεσμα να έχουμε μία ή δύο λιγότερες εκθέσεις ή να μην είναι τόσο εκτενείς οι εκθέσεις. Πρέπει μέχρι σε βάθος να φτάσουμε στη δράση μας και μέχρι τους αποδέκτες να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι ένα σημείο για την αναγνώριση επιπλέον του ευρωπαϊκού έργου που επιτελούμε εδώ προς όφελος των πολιτών και για καλύτερη ολοκλήρωση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ώστε οι κάτοικοι στις περιφέρειες, οι πολίτες να βοηθηθούν τελικά. Ως συντονίστρια για τους σοσιαλδημοκράτες θα ήθελα ένα πράγμα να τονίσω και να καταστήσω απόλυτα σαφές, ότι για είναι μια σαφέστατη θέση αυτή. Εμείς δεν θέλουμε όρους και προϋποθέσεις μακροοικονομικές να υπάρχουν στην πολιτική συνοχής. Εδώ πιστεύω ότι πρέπει να το πούμε διαζώσεις δυνατά και με ευκρινή τρόπο, με κάθε σαφήνεια. Δεν θέλουμε να υπάρξουν τέτοιοι περιορισμοί. Πρέπει να συζητηθούν βέβαια όλα αυτά τα πράγματα και πρέπει να, τα, ε, διαβουλευτούμε επ' αυτών ώστε να εξευρεθεί μια δυνατότητα να συνεργαστούμε αποτελεσματικά μαζί και να προαθούν αυτά. Θα έλεγα ότι για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων αυτά υπαρκούν από πλευράς μου. Και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν θα το καταφέρναμε να είχαμε μια πραγματικά έντονη συνεργασία σε βάθος ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Διότι η Δανέζικη Προεδρία είναι σε μια θέση που έχει σημασία κλειδιού για να προχωρήσουν όλα αυτά για την πολιτική συνοχή και για το χρονοδιάγραμμα που θέλουμε να τηρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κωνσταντσα εκ μέρου τη ομάδα Άλντε Μόνα Βαρεσκού. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον Υπουργό Βάμενε για την παρουσίασή του. Χαίρομαι που συμφωνούμε όλοι ότι η περιφερειακή ε, πολιτική και το ε, πολιετές ε, πλαίσιο είναι σημαντικό για την ανάκαμψη της Ευρώπης. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπαν οι δύο προλαλήσαντες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσθέσω ότι έχουμε ε, συνηθίσει σε ένα αποτελεσματικό μοντέλο ε, με την Πολωνική Προεδρία και περιμένουμε η Δανική Προεδρία να συνεργαστεί μαζί μας με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο, με το όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο, διότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις τις, ε, επόμενου επόμενους έξι μήνες για το νέο νομοθετικό πακέτο. Είναι λοιπόν ζωτικό για μας να ξέρουμε ότι θα μπορούμε να έχουμε διάλογο μαζί σας και ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα θέματα τα οποία ε, μας ενδιαφέρουν, που σχετίζονται με το νέο νομοθετικό πακέτο. Υπάρχουν Υπάρχει πληθώρα θεμάτων. Δεν πρόκειται να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, διότι ούτε η παρουσίασή σας, ούτε το έγγραφο εργασίας της Δανικής ε, Προεδρίας ε, δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες σχετικά με την περιφερειακή πολιτική. Αναφέρονται σε γενικότητες. Θα ήθελα όμως να σας θέσω δύο ερωτήματα. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την μακροαιρεσιμότητα. Όπως ακούσατε προηγουμένως, αμφιβάλλουμε για το γεγονός ότι υπάρχει, ότι είναι αποτελεσματικό να τιμωρούνται οι δικαιούχοι για τα σφάλματα των κυβερνήσεων. Και ένα άλλο θέμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ο περιορισμός του προϋπολογισμού. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η γνώμη σας για την απόφαση περικοπής από 3,8 σε 2,5 ε, του ΑΕΠ. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν, αλλά για την ώρα ε, θα ήθελα απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο επισημάνθηκε νομίζω και από τους τρεις συναδέλφους. Η Ιδανική Προεδρία επιθυμεί να έχει στενό διάλογο με το Κοινοβούλιο σχετικά με την πολιτική συνεχής. Ε, είναι γνωστό ότι οι πολιτικοί μακρηγορούν στις απαντήσεις. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω σύντομα, ταχύτατα, να πω ναι, το θέλουμε αυτό και περιμένουμε μια ισχυρή συνεργασία, μια αγαστή συνεργασία. Δεν θα υπάρχει άτυπη υπουργική συνάντηση για την συνοχή όπως έγινε με την Πολωνική Προεδρία. Όχι επειδή δεν πιστεύουμε ότι οι άτυπες συνεδριάσεις δεν είναι χρήσιμες, αλλά ε, Δανική Προεδρία θα έχει λιγότερες τέτοιες άτυπες συναντήσεις, όπως έγινε και σε άλλες προεδρίες. Αυτό που θα κάνουμε, θα έχουμε μερικές άλλες πρωτοβουλίες. Και ήθελα να πω ότι είμαστε ανοιχτοί για προτάσεις από το Κοινοβούλιο ε, και από αυτή την Επιτροπή για το πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία θα συμβούν την Άνοιξη είναι ότι και εμείς όπως και η Πολωνική Προεδρία θα έχουμε μια διάσκεψη για τα θέματα MFF όπου το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει βεβαίως. Θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο επικροτήθηκε από όλα τα κράτη-μέλη. Δεν πρόκειται να αναφέρω εδώ ονόματα, αλλά ε, δεν ξέρω αν όλα τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι είναι λαμπρή ιδέα να συνεχίσουμε αυτή την παράδειση. Αυτή είναι μια ένδειξη, ένα σημάδι της Δανική Προεδρίας ότι επιθυμεί να συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο. Θέλουμε να συνεχίσουμε μια τέτοια συνεργασία. Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι ότι θα έχουμε ε, συναντήσεις για την πολιτική συνοχή τον Απρίλιο και τον Ιούνιο. Και πριν από αυτές τις συναντήσεις όπως σε όλες τις συναντήσεις όπου θα συζητήσουμε το πλαίσιο MFFF, θα υπάρξουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον κύριο Λαμασούρ και άλλους όπου θα ασχοληθούμε με τα θέματα του πολιετούς πλαισίου, θα έχουμε στενή επαφή. Η ομάδα αυτή, συναδέλφων σας, ε, μας ρώτησαν αν θα μπορούσαμε να διευρύνουμε τις συναντήσεις αυτές εκ των προτέρων για να υπάρξει περισσότερος πραγματικός διάλογος ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, την Προεδρία και την Επιτροπή. Και η απάντηση της Προεδρίας ήταν ναι, μπορούμε να το κάνουμε, διότι θέλουμε καλή συνεργασία μεταξύ μας. Ο τρόπος λοιπόν εργασίας μας μπορεί να είναι κάπως διαφορετικός, αλλά ο σκοπός είναι ο ίδιος. Θα έλεγα επίσης ότι όλες οι καλές ιδέες είναι ευπρόσδεκτες και αν μπορώ να επανέλθω αργότερα στα θέματα αυτά θα ήμουν ευτυχής. Μπορούμε να συναντηθούμε με πρότυπο πιο άτυπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να επαναλάβω ότι θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά μαζί σας. Και σας το λέω και θέλουμε μια καλή συνεργασία, μια εταιρική σχέση και με αυτό το πνεύμα ήρθα εδώ σήμερα. Δεν είναι μόνο ε, ωραία λόγια τα οποία εκφράζω εδώ, ωραία λόγια της Δανικής Προεδρίας. Βεβαίω ο Λάμπερτ έθεσε τα ερωτήματα αυτά, τα θέματα αυτά και είπε επίση ότι είναι ουσιώδε ε, να ε, επιτύχουμε πρόοδο κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας και συμφωνούμε. Έχουμε μια προθεσμία η οποία είναι στην ατζέντα μας ότι το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο δεύτερο ήμιση του έτους αυτού, ακόμα και το θέμα της συνοχής. Για να καταστεί αυτό εφικτό θα χρειαστεί πάρα πολλές προσπάθειες της Δανικής Προεδρίας, αλλά επίσης και προσπάθειες του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Ούτω ώστε να μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα αντικείμενο διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο του Ιουνίου, βάσει του οποίου θα λάβουν χώρα διαπραγματεύσει στο δεύτερο ήμιση του έτους. Και αυτό θα πράξουμε Συμφωνώ λοιπόν με τα όσα είπατε, Λάμπερτ, για τα θέματα αυτά. Ξέρετε ότι αυτό το έχουμε πλήρως συνειδητοποιήσει. Αναφέρατε ε, ιδιαίτερα τις συναντήσεις και τις ε, διασκέψεις. Μου το είπατε και προσωπικά. Όταν τελειώσει αυτή η συνάντηση θα έρθω σε επαφή με τον Υπουργό που είναι υπεύθυνο για τη συνάντηση αυτή που δεν είμαι εγώ ίδιος ε, και θα του μεταφέρω τις απόψεις του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι θα αντιδράσει θετικά στο μήνυμα αυτό. Το δικό σας και άλλων συναδέλφων σας. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να προχωρήσουμε. Η Κωνσταντς είπε ότι είναι σημαντικό να έχουμε αυτή τη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Προεδρίας. Αλλά επίσης ανέφερε μερικά άλλα θέματα, παραμπτός χάρη, σχετικά με την αρχή της εταιρικής σχέσης των διαβουλεύσεων είναι κάτι το φυσικό και το σκόπιμο. Έρχομαι από μια χώρα που έχει παράδοση ως προς τις διαβουλεύσεις και για μένα αυτό είναι οφθαλμοφανές. Και θα ήθελα να συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο για το πώς θα μπορούσαμε να επιτύχουμε στο θέμα αυτό. Και εκτιμώ τις παρατηρήσεις που εκφράσατε εδώ σήμερα. Σχετικά με το θέμα της ε, μακροοικονομικής αιρεσιμότητας που τέθηκε τόσο από την Κωνσταντς όσο και από τη Ραμόνα. Βεβαίως πρόκειται για ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα, ας είμαστε ειλικρινείς. Ε, πρόκειται για ένα από τα δυσκολότερα θέματα που θα έχουμε επιτάπητος. Ξέρετε ότι θα συζητηθεί αυτό στο πλαίσιο ε, των φίλων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο στη ΚΑΚ όταν ε, θα, πρέπει να έχουμε στοιχεία τα οποία θα μεταφραστούν σε νομικές πράξεις. Δεν πιστεύω όμως ότι αυτό το μέρος της συζήτησης θα κλείσει κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας. Νομίζω ότι οι διχογνωμίες, οι διαφορετικές απόψεις και το εύρος, η σημασία των διαφόρων απόψεων στον τομέα αυτό θα παρατείνει τη συζήτηση αλλά σημειώνω τις απόψεις της Επιτροπής για το θέμα αυτό και θα διαβιβάσω το μήνυμά σας στο Συμβούλιο. Αλλά γνωρίζετε επίσης εδώ σε αυτή την αίθουσα ότι υπάρχουν διχογνωμίες και μέσα στο Συμβούλιο σχετικά με την προσέγγιση. Εν τέλει, ένας συμβιβασμός θα πρέπει να βρεθεί. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι θα διαβιβάσω το μήνυμά σας στο Συμβούλιο, διότι πρέπει να ξέρει ποια είναι η θέση αυτής της Επιτροπής. Επίσης, από τη Ραμόνα υπήρξε το θέμα ε, του κάπινγκ. Ε, ε, ναι, τονίσατε δικαίως ότι είναι από τα δυσκολότερα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια συζήτηση. Θα πρέπει όμως επίσης να πω ότι οι διαπραγματεύσεις για το MFF θα πρέπει να δείξουν αν η Κομισιόν έχει βρει τη σωστή ισορροπία. Διαφέρουν οι γνώμες μέσα στο Συμβούλιο. Αυτό δεν είναι μυστικό αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία έχει πλήρη συνείδηση της ιδιάζουσας κατάστασης επίσης ορισμένα κράτη-μέλη. Το γνωρίζουμε αυτό και πάλι είναι ένα από τα θέματα όπου εν τέλει τελικά πρέπει να βρεθεί ένα συμβιβασμό και θα μεταφέρω τις απόψεις της Επιτροπής αυτές στο Συμβούλιο και είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν πολύ για την άποψη των ομάδων στο Κοινοβούλιο είναι ένας από τους τομείς όπου θα συζητήσουμε μέχρι τέλους για να δούμε ποια είναι η δίκαιη λύση, η κατάλληλη λύση. Αυτό είναι έργο της Προεδρίας. Να μην φυστεί καμιά προσπάθειας για να φτάσει σε μια λύση που θα είναι αποδεκτή από τα κράτη-μέλη και από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Ευχαριστώ Γιάν Όλμπριχτ. Ευχαριστώ. Υπουργέ, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου. Πρόκειται για μια σαφέστατη δήλωση από πλευρά τη Δανέζικη Προεδρία, αυτή που δώσατε. Ότι θα συνεχίσετε δηλαδή την πορεία υποστήριξη ε, της πολιτική συνοχή ε, αφαιρετή. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλου μα διότι όχι μόνο η Προεδρία, αλλά βλέπουμε επίσης ε, και την θέση να εξειδικεύεται σε σχέση με σημαντικά κράτη-μέλη. Και ελπίζω ότι την ίδια θέση θα έχετε όπως τώρα και μετά τη Δανέζικη Προεδρία. Διότι οι υποχρεώσεις της Προεδρίας είναι πολύ συγκεκριμένες βέβαια. Ελπίζουμε στη συνέχεια βέβαια μετά την Προεδρία σας ότι θα συνεχίσετε να υιοθετείτε και να εκπροσωπείτε αυτές τις θέσεις. Περνώ τώρα σε κάποιες πιο συγκεκριμένες, πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις. Θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω το εξής. Πολύ περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα και γενική ερώτηση αυτή. Γενικά υπάρχει τάση είτε να ενδυναμώνεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε να μειώνεται, να συρρυκνώνεται η σπουδαιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή να διατηρείται ως έχει. Πιστεύω ότι πρόκειται για τις κατεντολήν πράξεις, εντεταλμένες πράξεις, κατεκπροσώπηση λοιπά. Δεν είναι μόνο το θέμα, θέματα που αφορούν τη δανέζικη κυβέρνηση. Είναι το πώς βλέπετε εσείς τα θέματα στο Συμβούλιο σήμερα. Βλέπουμε ότι ακολουθείται μια διαφορετική κατεύθυνση και υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ, τα οποία δεν εντάσσονται μέσα στον κανονισμό, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, Ποια είναι η θέση της Προεδρίας λοιπόν όσον αφορά περιβόητη, το περιβόητο μέσο για τις μεταφορές, transport facility, διότι αυτά τα κονδύλια βρίσκονται μέσα στο, στο πακέτο για τη συνοχή. Αν είναι μέσα σε αυτό υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αφαιρεθούν αυτά τα, κίνδυνα, τα κονδύλια από τις ε, χώρες ε, συνοχής, 10 δισεκατομμύρια. Δεν πρόκειται, δεν πρόκειται μόνο για την αφαίρεση κονδυλίων, αλλά όταν τα παίρνουν, τα αφαιρούν, και μετά δίνονται στην αποκαλού, αποκαλούμενες οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Τι γίνεται εδώ όμω με την επιμερισμένη διαχείριση, με την κοινή διαχείριση. Δεν θα είναι αυτή αυτή η αρμοδιότητα θα είναι αρμοδιότητα κάποιου, κάποιων στις ε, Βρυξέλλες με μια δημόσια προσφορά, με, με προσφορές που θα υποβληθούν. Σε μια τέτοια διαδικασία είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό να προκαθορίσουμε τα κονδύλια αυτά που θα διατεθούν. Να μην τα αφαιρέσουμε από τις χώρες συνοχής. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για όλε τι χώρε συνοχή. Και θέλω να σα το πω, να σα ενημερώσω ότι έχουμε συναντήσει εδώ στο κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου και ακούμε από την Γενική Διεύθυνση για Περιφερειακά Θέματα που παρίσταται ότι θα αφαιρεθούν αυτά τα κονδύλια. Έχουμε τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών που μα λέει όχι, θα δοθούν αυτά τα χρήματα, δεν θα αφαιρεθούν. Είμαστε λοιπόν, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να δοθούν τα πρόσθετα 10 εκατομμύρια στι χώρε συνοχή. Ξέρουμε όμω τι γίνεται. Δεν δίνονται αυτά, αφαιρούνται και τα προβλήματα βρίσκονται στις λεπτομέρειες. Επιμερισμένη διαχείριση, σταθερή, σταθεροποιημένη διαχείριση. Δεν είναι μόνο, τα πόσα, δεν είναι μόνο το θέμα περί τίνων κονδυλίων πρόκειται. Και έχουμε και το ε, ESF, δηλαδή τι θα έχουμε καθορισμένα κονδύλια στο σύνολο του πακέτου. Για παράδειγμα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες σε 25, κατά 25% ή στις ε, κατά 40% χώρες. Ή θα είμαστε πιο ευέλικτοι και θα αφήσουμε τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν που βρίσκονται εκτό κανονισμού. Είναι όμω σημαντικότατα για του ίδιου του κανονισμού. Διότι χωρί να επιληθούν τα προβλήματα για το μέσο για τι μεταφορέ και το ESF θα έχουμε προβλήματα. Θα έχουμε πολύ δυσχερή κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που αφορά τον ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο, δεύτερο το διαβόητο θέμα για το μέσο αυτό και την διευκόλυνση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι στις συζητήσεις ε, ε, από πλευράς ε, της Επιτροπής θα υπάρχει δυνατότητα να προσέλθετε και εσείς ως συγητής και να συζητηθούν αυτά στην Κοπενχάγη, να συνεργαστούμε, να έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τις δανέζικες αρχές να συζητηθούν στην Κοπενχάγη για τους κανονισμούς. Ελπίζουμε ότι θα, είναι, θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Εσείς έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από μια ώρα ξεκινήσαμε μια συζήτηση για ένα εξειδικευμένο θέμα. Όμως, φαίνεται ότι εδώ δεν υπάρχουν, ε, από ό,τι φαίνεται, κάποια προβλήματα στο Συμβούλιο για το μηχανισμό επιμερισμού για τα κράτη-μέλη που έχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση των σχεδίων και προγραμμάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει κοινή συνένεση στην Επιτροπή Περιφερεια... από την ε, Ρέτζι και στην... Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετηθεί ταχύτερη διαδικασία, επισπεσμένα και σε σχέση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσουμε. Όμως φαίνεται από την άλλη πλευρά ότι κάποιοι στο Συμβούλιο δεν συμφωνούν, κάποιος φταίει και κάτι γίνεται και δεν προχωράμε από το Δεκέμβριο και από την τελευταία συνάντηση της ομάδας εργασίας δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. Τι γίνεται, μπορείτε να μας επεξηγήσετε περισσότερο με κάποιες λεπτομέρειες γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί η πρόταση αυτή έχει τροχοπεδηθεί. Είναι μια κατεπήγοντος χαρακτήρα πρόταση και αυτός ο μηχανισμός έχει μεγάλη σημασία και σπουδαιότητα για την Ελλάδα και πρέπει να βοηθήσουμε το δυνατόν ταχύτερα. Αλλά και για άλλες χώρες είναι σημαντικός. Αυτό λοιπόν τώρα και προσωπικά από πλευρά μου. Αναφέρατε τη διαδικασία για την οδηγία δημοσίων προμηθειών, θα μπορούσατε, δημοσίων αγορών. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά. Αναμένουμε εμείς αυτή την πρόταση και ακούμε ότι δεν έχει γίνει και τίποτα. Αν υπάρχει κάποια ιδέα ή άποψη για το χρονοδιάγραμμα και πώς μπορεί να προχωρήσει, να μας τα πείτε παρακαλώ. Κοίταξε από παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την εξαιρετική σας εισήγηση. Όπως αναφέρθηκε από τους συναδέλφους επανειλημμένα, από πλευράς ε, και της Πολωνικής ε, Προεδρίας είχαμε συνηθίσει μια σφιχτή αποτελεσματική Προεδρία. Είχε προτεραιότητα αυτό το θέμα για τους Πολωνούς, για την Πολωνική Προεδρία. Και για την Προεδρία της Δανίας ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί και να δοθεί συνέχεια σε αυτό από πλευράς ε, των κονδυλίων κατά τους επόμενους έξι μήνες για την πολιτική συνοχή. Στις συζητήσεις αναφέρθηκαν πολύ σημαντικά θέματα στις παρεμβάσεις. Κάποια σχόλια και ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Για παράδειγμα, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντικό εδώ. Έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα να δούμε οι περιφέρειες να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτές τις συμφωνίες συνεργασίας, ώστε η συνεργασία και οι δράσεις να ξεκινήσουν στο περιφερειακό επίπεδο και να συνεχιστούν στο κρατικό επίπεδο. Φοβούνται όμως πολύ. Υπάρχουν φόβοι και επιφυλάξεις ότι θα επικεντρωθούμε όλο και περισσότερο στις κρατικές κυβερνήσεις, κρατικές αρχές για τη διάθεση αυτών των κονδυλίων και τις δικές τους δράσεις και όχι τόσο στις περιφέρειες. Πρέπει να λυθούν τα βήματα και διαβήματα προς την ορθή κατεύθυνση. Μία ερώτηση θα ήθελα να διατυπώσω προ τον Υπουργό, διότι ανέφερε ότι όσον αφορά την απλούστευση έχετε προχωρήσει λέει, λίγο πιο πέρα και έχετε συζητήσει περισσότερο τα θέματα αυτά της απλούστευσης. Ποια είναι τα συγκεκριμένα χειροπιαστά αυτά ε, μέτρα ω προτάσει που υπάρχουν τώρα διότι όσον αφορά την καταποκοπή ε, ε, καταβολή ποσών, ε, πώς θα προχωρήσετε για την απλούστευση. Πρέπει να θυμόμαστε όμως πάντα ότι στο επίπεδο των κρατών μελών το γραφειοκρατικό βάρος είναι διαφορετικό, υπάρχουν σημαντικές διαφορές και εδώ πάλι ελπίζω ότι θα υπάρχει μια πιο συνεκτική, με μεγαλύτερη συνοχή προσέγγιση όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή από τα κράτη-μέλη όλων αυτών. Και μετά για, τη μεταφορά, για τις μεταφορές και τις περιφέρειες. Έχετε κάποια αριθμητικά μεγέθη. Πώς όλα αυτά, ποιες επιπτώσεις θα έχουν στη συνολική πολιτική και ποιες συζητήσεις και ποια αποτελέσματα σημειώνονται. Αυτό και πάλι θα είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα όσον αφορά την μελλοντική νομοθεσία, το μελλοντικό νομοθετικό έργο. Επιπλέον κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά ως τον ρόλο που είχα αναλάβει ε, για την εισήγηση που μου είχε ανατεθεί, θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία, την δράση στο περιφερειακό επίπεδο και το νομοθετικό έργο. Υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν εξεταστεί, έχουν συζητηθεί. Πώ εσεί ω Προεδρία θα επικεντρωθείτε σε αυτό. Και όσον αφορά τα δημοσιονομικά θέματα, το προπολογισμό και τα κονδύλια, θα είσαστε υπέρ του το επίπεδο προπολογισμού να είναι στο 3,5 όπω αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Υπουργέ, εσεί έχετε τον λόγο τώρα. Σα ευχαριστώ πολύ. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφέρω το εξή. Να στραφώ στον Γιάν και να του πω, ο οποίο ανέφερε προηγούμενα ότι αν η δανέζικη θέση θα είναι ακριβώς η ίδια μετά τη δανέζικη προεδρία ή όχι. Η ίδια με εκείνη που είχε η δανέζικη προεδρία κατά την διάρκεια τη προεδρίας τη. Προσωπικά τον φίλο Νικολάη για τα ευρωπαϊκά θέματα άκουσα ότι μετά την Προεδρία που είχε αναλάβει η Πολωνία τώρα πλέον εφ' εξής θα εργαζόταν αποκλειστικά για πολωνικά συμφέροντα αναγνωρίζοντας έτσι ρητά το γεγονός ότι ο ρόλος ε, της Προεδρίας μιας χώρας είναι κάτι το ξεχωριστό και εξαιρετικό. Και γι' αυτό είναι σημαντικό για μένα να πω ότι εγώ εκπροσωπώ ως Προεδρεύω του Συμβουλίου 27, 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο τη Δανία. Άσχετα από τις επιμέρους εθνικές θέσεις, εγώ δεν τοποθετούμε εδώ εξ ονόματος της δανέζικης κυβέρνησης αλλά Ομιλώ εξ ονόματο τη Δανέζικης Προεδρία του Συμβουλίου. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε μια με ανοιχτό πνεύμα Προεδρία, με επικοδομητικό πνεύμα Προεδρία του Συμβουλίου. Και θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα κοινό πλαίσιο στο οποίο θα αντανακλώνει τα συμφέροντα και των 27 κρατών μελών. Ελπίζω ότι θα βρείτε λοιπόν και την Δανέζικη Προεδρία όπως την Πολωνική Προεδρία. Μια Προεδρία με πολύ ανοιχτό πνεύμα, με επικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας. Αυτός είναι ο στόχος ε, και η στοχοθέτηση. Αυτή πάντα ήταν και η θέση, η τοποθέτηση της Δανίας και ως εθνικής κυβέρνησης πριν από την Προεδρία αλλά και μετά Προσπάθεια δηλαδή να δώσουμε αυτή την ε, γραμμή και πορεία στην Κυπριακή κυβέρνηση στη συνέχεια, Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου. Με χαρά μπορώ να το αναφέρω λοιπόν αυτό ότι με αυτή τη βάση εργαζόμαστε. Ερώτηση που διατυπώσατε σε σχέση με το Connecting Europe, το μέσο διευκόλυνσης ε, σύνδεσης ε, μεταφορικά της, και των μεταφορών της Ευρώπης. Πρώτον, θα πρέπει να διασφαλιστεί αυτή η πρωτοβουλία. Και δεύτερον, να προσπαθήσουμε αυτά τα δισεκατομμύρια, όπως λέτε, ευρώ σε σχέση με την ε, συνοχή για την να χρησιμοποιηθούν τα, ε, ή, τα σχέδια της ε, διασύνδεσης της Ευρώπης. Θέλουμε φυσικά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση δικτύων. Όμως δεν υπάρχει κάποιο μυστικό εδώ ότι αν αυτά θα κονδύνε, θα προέρχονται από το πακέτο για τη συνοχή ή όχι και θα μπορούσε να είναι αυτό το ποσό μεγαλύτερο, μικρότερο. Πολλέ συζητήσει διεξάγονται και πολλά λέγονται. Ε, αυτό λοιπόν πρέπει να το διαπραγματευτούμε. Θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση. Και εδώ πάλι μπορείτε να βρείτε διαφορετικέ απόψει στα μέλη του Συμβουλίου στι τοποθετήσει του. Γι' αυτό συνειδητοποιώ, έχω συνειδητοποιήσει απόλυτα το θέμα η Προεδρία έχει συνειδητοποιήσει και γνωρίζει πολύ καλά αυτό το θέμα και ευελπιστώ πρέπει να πω με κάθε τρόπο ότι η δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή όπως και το Ευρωκοινοβούλιο στο σύνολό του θα γνωρίζουν τα τεκτενόμενα και θα δράσουν συνειδητά. Έχω όμως καλά σημειώσει τα όσα είπατε για τον προκαθορισμό κονδυλίων από πλευράς ESF. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και πάλι εδώ δεν μπορώ να δώσω κάποιες τελικές καθοριστικές τοποθετήσεις στις δηλώσεις μου. Απλώς να πω ότι αυτό θα είναι ένα από τα ζωτική σημασία θέματα στα οποία πρέπει να εξευρεθεί και γι' αυτό μια λύση τους επόμενους μήνες. Και βλέπουμε ότι έχουμε αυτά τα θέματα τα οποία τίθενται επί από την κοινοβουλευτική σας επιτροπή σήμερα. Δεν είναι κάτι όμως για αυτά στα οποία έχουμε την λύση κομμένη και ραμμένη έτοιμη σήμερα. Αν ήταν εύκολο θα ήταν γνωστό αυτό, αλλά δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε φυσικά να αποκρισταλωθεί μια άποψη στο Συμβούλιο για αυτά τα θέματα και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε έναν πολύ επικοδομητικό, δημιουργικό διάλογο με τη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και τους Ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο ώστε όπως είπαμε και στην Κοπενχάγη να προσέλθετε να μας επισκεφτείτε το καλωσορίζω αυτό αν μπορεί να γίνει με ιδιαίτερη χαρά θα έβλεπα μια τέτοια αποστολή σας ώστε να συντονιστεί έτσι αυτή η αποστολή σας με τη Δανέζικη Προεδρία ώστε να έχουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις να σας ενημερώσουμε και να βοηθήσετε να παρακολουθήσετε τα προγράμματα εκείνα και σχέδια που μπορούν να είναι υποφελή και ή δυνατόν να είναι στη διάθεσή σας και ο Υπουργός Εξωτερικών και να υπάρχει δυνατότητα και να έρθουμε και εμείς σε εσάς, αλλά εσείς να έρθετε και εσείς στην Κοπεχάγη και να προσπαθήσουμε να δούμε αν όλα αυτά μπορούν να στεφτούν με επιτυχία ως εγχείρημα προς το συμφέρον αυτό όλων μας πιστεύω. Τώρα το ερώτημα που διατυπώθηκε για την θεματολογική επικέντρωση, thematic concentration, είναι ένα δύσκολο, δυσχερές θέμα αυτό. Και από πλευρά του Συμβουλίου δεν βρήκαμε ακόμα την τελική, ας το πω έτσι, κατεύθυνση που να μας ενώνει σε μια σύμφωνη πορεία όλους μας. Συνεχίζουμε όμω ω ε, Δανέζικη Προεδρία για να το πετύχουμε αυτό. Ρωτήθηκε για το μέσο επιμερισμού κινδύνων για τις δράσεις μας. Είναι μια σχετικά νέα βέβαια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο Συμβούλιο είχαμε μια παρουσίαση και μια πρώτη συζήτηση τη πρόταση αυτή κατά τη διάρκεια της Πολωνικής προεδρία, βέβαια. Και η στρατηγική τη Δανέζικη Προεδρία είναι να διαβουλευτούμε και να προετοιμάσουμε το χαρτοφυλάκιο σε βάθος, ώστε να έχει οριμάσει. Όταν θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για αυτές τις προτάσεις να έχουν οριμάσει κάποια πράγματα. Προ αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σύμφωνη γνώμη με την Προεδρία θα διεξαγάγει ήδη αύριο ένα τεχνική φύσεως, τεχνικού χαρακτήρα σεμινάριο και εγώ θεωρώ ότι ο κύριος στόχος αυτών των ε, ε, προτάσεων είναι να μπορέσει να προαχθεί ο επιμερισμός κινδύνου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα συναφή όργανα όταν θα δίνονται δάνεια ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση για τέτοια σχέδια. Οι κύριες αρχηριότερες αρχές γίνονται κατανοητές βέβαια, αλλά οι λεπτομέρειες πρέπει να εξειδικευτούν και να αποκρισταλωθούν. Συνεχίζεται η δουλειά προς αυτήν την κατεύθυνση. Συμφωνώ μαζί σας, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα ποιότητα και ο χρόνο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο φίλο, όπω είπατε εσεί μπορεί να είναι φίλο. ο χρόνο μπορεί να είναι φίλο. Πολλέ φορές ε, δεν υπάρχει πολλής χρόνος, αλλά έχει κανεί πολλούς φίλους. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε. Η Προεδρία, εν πάση περιπτώσει, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τη. Να αναλάβει εκείνα τα βήματα και διαβήματα για να προχωρήσει. Για το θέμα των δημόσιων αγορών και προμηθειών θα πρέπει να επανέλθουμε στη συνέχεια να ε, όταν θα έχουμε την ημερομηνία να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες όταν θα έχουν οριμάσει κάποια πράγματα. Εσείς στη συνέχεια αναφέρατε πολλά σημαντικά θέματα, Ευρωβουλευτά, και αν δεν είμαι και σε θέση να τα απαντήσω όλα όσα αναφέρατε σήμερα, ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να επανέλθουμε να τα συζητήσουμε περαιτέρω και να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Για την απλούστευση είναι ένα δυσχερές ακαθόδες θέμα όπως αναφέρατε συζητούμε τα ποσοστά τα οποία αφορώνται εδώ έχουν σημειωθεί αυτά την Επιτροπή. Η πραγματική πρόοδος όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει ακόμα να επιτευχθεί. Θέλουμε να επιτευχθεί για να υπάρχει περαιτέρω απλούστευση όπου είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Πρέπει να είναι πολύ σημαντικό βέβαια ο στόχος το ότι οι κανόνες και οι κανονισμοί θα διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι το δυνατόν πιο εύληπτοι και πιο ε, ευσύνοπτοι ενώ ταυτόχρονα θα είναι αποτελεσματική. Και μια γενικότερη συζήτηση εδώ ε, θα πρέπει να εμπλέξει αυτά τα θέματα. Είναι μια από τις συζητήσεις που είχαμε και γενικότερα για την πολιτική συνοχή μεταξύ του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τότε δηλαδή δεν θέλουμε να έχουμε όλο και περισσότερο γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, γραφειοκρατικό βάρος. Θέλουμε να απλουστευτεί το γραφειοκρατικό βάρος και η γραφειοκρατική δυσκολία να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με πιο απλό, ε, εύκολο, πιο θα έλεγα εύκολο να ακολουθηθεί σε διεργασίες και διαδικασίες τρόπο, με λιγότερη γραφειοκρατική επιβάρηση. Κάνετε επίσης λόγο και για μια μεταβατική προσωρινή περίοδο για τις ε, χώρες υποστήριξης. Και αυτό θα είναι μέρος των διαπραγματεύσεων. Όπως γνωρίζετε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτει δύο διαφορετικές ε, περιπτώσεις. Πρώην περιοχές ε, σύνοχης, σύγκλησης για την η μία περίοδο επταετή και δεύτερον άλλες περιοχές με ΑΕΠ μεταξύ 75 και 90 του μέσου όρου της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ώστε να μπορέσουν ε, να ενισχυθούν ανάλογα με την θέση που, στην οποία βρίσκονται στις, μεταξύ των περιφερειών. Αυτό συνδέεται με το θέμα ποιος πληρώνει τι για ποιον. Και δεν μας εκπλήσει φυσικά, δεν πρέπει να εκπλήσει κανένα ότι διήστανται οι απόψεις και υπάρχουν διαφορές θα πρέπει να ληφθούν τέτοιε αποφάσεις ώστε να εξισορροπούνται οι ανάγκες των περιφερειών με τα μέσα που είναι διαθέσιμα και τις δυνατότητες. Και πάλι πιστεύω ότι αυτό το τμήμα θα μπορέσει να επιληθεί ως μέρος ενός συμβιβασμού μέσα στο πλαίσιο των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών. Δεν είμαι σε θέση να δώσω καθοριστική απάντηση ακόμη σήμερα. Όμως αυτό πρέπει να δούμε ποια τελική έκβαση θα ε, πάρει. Αναφερθήκατε και στην συνεργασία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, περιφερειακά, διαμεθοριακή συνεργασία και τα συναφή σε σχέση με τα άλλα δημοσιονομικά μέσα της ε, Ένωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δεύτερο σκέλος. Ακολουθούμε το πολωνικό πρότυπο το να υπάρξουν κάποιες ε, δυνατότητες ε, να προχωρήσουμε απλουστεύοντας τα θέματα όσον αφορά και τη διαχείριση και τα ζητήματα ελέγχου και κατά τη διάρκεια της Δανέσκης Προεδρίας σε σχέση με τα άλλα μέσα τα οποία έχουν σχεδιαστεί γνωρίζω τις τα μελήματα και τις ανησυχίες σας όσον αφορά το, μέλος, το μέσο γειτονία και την δυνατότητα δραστηριοποίησης όσον αφορά την ανάπτυξη των περιφερειών. Εδώ θα πρέπει να συνδέεται αυτό με το δικαίωμα ανάληψης ιδίας πρωτοβουλία ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φοβούμε ότι αυτή η ολοκλήρωση σε όλες τις πτυχές δεν έχει εγγραφεί στην ημερησία διατάξη. Από την άλλη πλευρά η εργασία με το μέσο γειτονία, το ENPI, στα εξωτερικά σύνορα έχει και αυτό τη σημασία του. Ελπίζω λοιπόν ότι μαζί με τα άλλα θέματα που αναφέρατε ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στη συνέχεια ως Προεδρία σε εσά να σας ενημερώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και Ιωάνν Ιωκαμ Τέλλορ Βίκτορ Μπορσινάν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Δανό Υπουργό για το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε. Έχω δύο εξειδικευμένες ερωτήσεις, οι άλλες απαντήθηκαν. Ε, το σας ευχαριστούμε που προσπαθείτε να βρείτε έναν κοινό δρόμο για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους έξι επόμενους μήνες. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας ε, διότι τα κρατη θα μειώσουν, θα περικόψουν ε, τις δημόσιες δαπάνες λόγω κρίσης. Πώς η Ιδανική Προεδρία θα ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τους νέους. Η γνώμη μας ε, είναι ότι η πολιτική συνοχή θα έπρεπε να συμβάλλει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κυρίως για τους νέους. Έχουμε έναν μέσο όρο περίπου 21% για τους νέους ανεργίας και χώρες όπως η Ισπανία έχουν 40% ανεργίας των νέων. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας κυρίως για τους νέους. Και πώς και αυτό από την άποψη των διαπραγματεύσεων για την πολιτική συνοχή θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι. Δεύτερον, ε, ποια είναι η άποψη της Δανικής Προεδρίας ως προς μια πράσινη Ευρώπη. Πώς σε μια πιο πράσινη Ευρώπη μπορούμε να ε, προωθήσουμε ορισμένα μέσα στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και ποιε είναι οι σχέσεις ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και τις άλλες τομεακές πολιτικές. Ναι, σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς πολύ Υπουργέ που ήρθατε εδώ ενώπιον μας. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για το ότι από τη θέση ενός κράτους μέλους που είναι καθαρός εισφορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς επιφύλαξη υποστηρίζεται την πολιτική συνοχή και τη θεωρείται ένα από τα σημαντικά πολιτικά πεδία στα οποία πρέπει να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προηγούμενα υπήρχαν κάποιε ανησυχίε, βέβαια όσον αφορά τη Δανέζικη Προεδρία όταν θα ερχόταν η ώρα τη να αναλάβει τη σκητσάλη από του Πολωνούς αν θα άλλαζε κάποια κέντρα βάρου ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ που αντιμετωπίσατε αυτέ τι ανησυχίε και η πολιτική συνοχή και η διαρθρωτική πολιτική θα προαχθεί και θα τονωθεί από τη δική σα Προεδρία όπω είπατε και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Αυτά που ανέφεραν οι συνάδελφοι δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα από όσε υπάρχουν απαντήσεις διαθέσιμες. Και το πρόβλημα του χρόνου είναι φυσικά ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Ιδιαίτερα σε αυτή την Δανέζικη Προεδρία του Συμβουλίου θα πρέπει να τεθούν τα ορόσημα, διότι το 2014 δεν απέχει πια τόσο από την, το σημερινό έτος. Και αν θέλουμε τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν την πολιτική συνοχή και στα διαρθρωτικά, θα εξαρτώνται φυσικά από το να, γνωρίζουν, να γνωρίσουν σε ποια βάση θα μπορούν να δράσουν Δηλαδή τα λειτουργικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ποια κατεύθυνση θα πορεύονται με τις αναγκαίες συμβάσεις και συμφωνίες και την υποστήριξη για τη διαφορετική πολιτική που θα διασφαλιστεί από το Συμβούλιο. Γι' αυτό εξαρτάται από τη δική σας προεδρία σε μεγάλο βαθμό και από τη δική σας ικανότητα στις διαπραγματεύσεις να τεθούν αυτές οι προϋποθέσεις και οι όροι ώστε να ευδοκιμήσουν αυτοί οι στόχοι. Τον μερικό τομέα των διασυνοριακών συνεργασιών θα ήθελα να θίξω τώρα. Οι συνάδελφοι είπαν πιο πριν ότι πολλά πράγματα απαιτούν μια καλύτερη, πιο ευσύνοπτη, ας το πω έτσι, λειτουργία. Αλλά και τα αναγκαία χρηματοοικονομικά μέσα πρέπει να διατεθούν όπως είναι αναγκαίο για να λειτουργήσουν αυτά τα σχέδια. Αναφέρατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι έχει την υποχρέωση να αναλάβει πρωτοβουλίε από πλευρά τη. Όμω, βλέπω και παρατηρώ ότι ακριβώ στο επίπεδο πολλών κρατών μελών υπάρχουν διαφορετικέ απόψει για αυτά τα θέματα. Θα σα παρακαλούσα λοιπόν θερμά γι' αυτό εσείς Υπουργέ Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, στο επίπεδο των κρατών μελών, να δράσετε ώστε να τοποθετηθείτε με σαφήνεια για αυτά τα θέματα. Και τα ίδια ενισχύει μέσα που λειτουργούν στα πολιτικά πεδία και στα νομικά πλαίσια για τον, ε, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, περιφερειακής συνεργασίας να δράσουμε και να προχωρήσουμε. Τη διαμεθοριακή συνεργασία τη θεωρώ πυρήνα, καρδιά της ε, συνεργασίας μας στο περιφερειακό επίπεδο. φορές βρίσκονται οι περιφέρειες λιγότερο ανεπτυγμένε περιφερειέ τη ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές οι μεθοριακές περιοχές. Πρέπει η Ευρώπη να ολοκληρωθεί, να προσεγγίσει μια περιφέρεια την άλλη και να ανέβει το επίπεδο. Η Δανία, όπως και 7 άλλε περαιτέρω χώρες, βρίσκονται στις μακροπεριφέρειες της Ευρώπης, δηλαδή τη στρατηγική για τις χώρες της Βαλτικής, μία από τις λίγες αυτές εγκεκριμένες ομάδες και στη Σουηδία αυτή η στρατηγική εγκρίθηκε και αναμένουν πολύ, πολλά πράγματα, όχι μόνο όσον αφορά τη Βαλτική θάλασσα, συνολικά, αλλά ποια συνέχεια θα δοθεί και ποιο μέλλον θα υπάρξει για άλλες μακροπεριφέρειες, μεγαλύτερες δηλαδή ενώσεις χωρών σε μακροπεριφέρειες στην Ευρώπη. Εξαρτώνται αυτά από τη δική σας διαρθρωτική πολιτική. Έχουμε το κέντρο μεταξύ Στοκχόλμης, Κοπενχάγης και Όσλο στις σκανδιναβικέ χώρες. Έχουμε όμως και άλλες χώρες που εξαρτώνται ιδιαίτερα από τη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Thank you very much Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ Βάμεν για την προθυμία σας, το ανοιχτό σας πνεύμα και τις πλήρεις απαντήσεις που μας δίνετε. Μια παρατήρηση. Μπορώ να προσθέσω νέες ερωτήσεις και ανησυχίες σχετικά με το πρόγραμμα Connecting Europe, διασυνδέοντας την Ευρώπη. Αλλά δεν είναι η στιγμή να διευρύνουμε τη συζήτηση. δεύτερη ερώτηση ε, σχετικά με την επίδοση ε, υπάρχει ένα θέμα όπου έχουμε διχογνωμίες όχι μόνο μέσα στην Επιτροπή αλλά και μέσα ε, στο Συμβούλιο για την Performance Reserve. Ποια είναι η θέση του της Δανικής Προεδρίας για την εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά και ίσως το άνοιγμα του, Ταμείου Συνοχής για επιδότηση τέτοιων προσπαθειών. Είχα ουσιαστικές συζητήσεις με τις Επιτρόπους Ποτότσκιν και Χέντεγκαρντ είναι θετική και τον Μάρτιο θα οργανώσουμε ένα συνέδριο και είμαι πεπισμένος ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Ποια είναι η ιδανική θέση. Και η τελευταία ερώτηση. Ξέρω πολύ καλά ότι τον Μάρτιο ο Επίτροπος Ποτόσνικ θα ανοίξει τις συζητήσεις για νέες οδηγίες και αξιολόγηση ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου και στρατηγικού αντικτύπου. Ε, τι, ποια είναι η θέση της Δανικής Προεδρίας για τα σημαντικά αυτά θέματα, διότι είναι ζωτικό να δούμε τις απαντήσεις. Αν θέλουμε να συνδέσουμε την δυνατότητα πρόσβαση στο Ταμείο Συνεχής στις περιπτώσεις όπου ο ρηπαίνων δεν πληρώνει, διότι αυτή θα είναι η τελευταία δυνατότητα, τελευταία δυνατότητα και όχι μία τακτική δυνατότητα. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση από μέλη της Επιτροπής. Α, όχι, όχι, υπάρχει ακόμα. Κάποιος που θέλει να λάβει το λόγο. Α, απλώς θα ήθελα να πω κάτι. Ήταν μεγάλη προσπάθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για να έχουμε πολύ ε, καλούς ε, διερμηνείς για την δανέζικη γλώσσα. Ελπίζω να μας πείτε κάτι στα δανέζικα. Για την ώρα, όσοι Φατούρα. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Έχω τρεις ερωτήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί για το Ταμείο Αλληλεγγύης, ποια είναι η κατάσταση. Δεύτερον, εμείς στην Επιτροπή Ρέτζη συζητούμε πάρα πολύ ε, για την επικουρικότητα ε, με την διασύνδεση με τους πολίτες, με την τοπική αυτοδιοίκηση, αποκέντρωση, πώς να είμαστε πιο κοντά στους πολίτες όταν λαμβάνουμε αποφάσεις και ο Υπουργός δεν τόνισε αρκετά το ρόλο των περιφερειών σχετικά με το νέο πακέτο που συζητούμε. Πώς λοιπόν εσείς αντιλαμβάνεστε το ρόλο των περιφερειών θα ενισχυθεί στην επόμενη περίοδο. Ε, και η τρίτη ερώτηση πολύ σύντομη. Οι συζητήσεις μας εστιάζονται στο μελλοντικό νομοθετικό πακέτο, όμως παρόλα αυτά θα ήθελα τη γνώμη σας για την σημερινή κατάσταση. Η Ευρώπη φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Η οικονομική ανάπτυξη είναι στάσιμη στην Ευρωζώνη και εκτός της Ευρωζώνης. Και θα ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με την κατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη τώρα. Θα ήθελα να αρχίζοντας με απαντήσεις για τις τελευταίες ερωτήσεις ε, που σχετίζονται με τα όσα ρώτησε ο Πίτρου, πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θα ήθελα να πω ότι η βασική προτεραιότητα της Δανικής Προεδρίας είναι να ξαναρχίσει να λειτουργεί καλά και να δουλεύει καλά η Ευρώπη. Υποστηρίζουμε τα μέτρα λιτότητας, αλλά δεν μπορούν τα μέτρα αυτά να είναι μόνα τους. Θα πρέπει να τα συνοδεύσουμε με πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν τις δυνατότητες οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης της Ευρώπης και που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η Δανική Προεδρία έχει δεσμευθεί ε, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας ε, για τους νέους στην Ισπανία όπου 45% των νέων δεν έχουν δουλειά, αυτό είναι κάτι που έχει επιπτώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν ιδιαίτερη υποχρέωση να δώσουμε απαντήσεις στους νέους. Να ανταποκριθούμε. Νομίζω ότι η μεταρρύθμιση της ενίας αγοράς θα συμβάλλει σημαντικά στο θέμα αυτό. Τα πρώτα δέκα χρόνια είχαμε 2.500.000 θέσεις εργασίας. Πιστεύουμε επίσης ότι τόσο για το Ταμείο Συνοχής και τα ταμεία του MFF γενικά, ότι θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι κάθε ευρώ που ξοδεύεται θα δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση. Αυτό είναι ζωτικό. Έχουμε πλήρη συνείδηση του γεγονότος αυτού και κάθε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας θα έχουμε θα αποδώσουμε ιδιαίτερη ε, σημασία στην αναμόρφωση της ενίας αγοράς ε, κατά τη διάρκεια των 5-6 μηνών που θα έχουμε ως Προεδρία θα εστιαστούμε στο θέμα αυτό και για το δεύτερο θέμα σχετικά με την πράσινη ατζέντα ξέρω ότι υπάρχουν μερικοί στην Ευρώπη που λένε ότι με την πράσινη θα πρέπει να έχουμε περισσότερη πράσινη βιομηχανία, πράσινη οικονομία. Αυτό βεβαίω μπορεί να επιβαρύνει άλλους τομεί. Νομίζω ότι ο σωστό τρόπος να τα βλέπει κανείς τα πράγματα είναι απλό. Οι θέσει εργασία θα δημιουργηθούν παγκοσμίω με την πράσινη οικονομία. Το θέμα δεν είναι αν θα δημιουργηθούν, το θέμα είναι θα δημιουργηθούν εδώ στην Ευρώπη ή θα δημιουργηθούν στις Ηνωμένε Πολιτείε, στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Στις άλλες χώρες BRIC. Εμείς δεν θα αφιστούμε καμιάς προσπάθειας για να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες που θα μπορούν να προωθήσουν αυτή την ατζέντα, διότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα προκαλέσει ανάπτυξη έχουμε δεσμευθεί για το θέμα αυτό. Ο Ιόκιμ επεσήμανε ένα θέμα και είπε ποια είναι η άποψή μας για την μακροοικονομική περιφερειακή πολιτική. Έχουμε τη Βαλτική Πρωτοβουλία, αλλά έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να ανακύψουν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό οι στρατηγικές να αναπτυχθούν μέσα στα ήδη φυστάμενα πλαίσια. Δεν θα υπάρξει λοιπόν νέα νομοθεσία, νέες δομές χρηματοδότησης. Πώς θα μπορούμε καλύτερα να εξασφαλίσουμε με τα σημερινά ε, ταμεία μέχρι το 20 να επιτύχουμε μέσα στο πλαίσιο αυτό δεν μας φαίνεται παράλογο να ε, δούμε ε, ε, στη διαδικασία του προγραμματισμού ε, τα μακροοικονομικά και θα ήθελα να συγχαρώ την Κομισιόν για αυτό που νομίζω ότι είναι καλή πρόταση αυτή που υπέβαλε. Είναι μια καλή πρόταση. Οι ε, μακροπεριφερειακές στρατηγικές είναι σημαντικό εργαλείο για την συνοχή ανάμεσα σε διάφορες χώρες και περιφέρειες. Αν διευκολύνουμε ε, τις ισχυρές υποδομές και την πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη, οι, μακρο, οι μακροοικονομικές στρατηγικές θα είναι προστιθέμενη αξία. Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι αυτά που κάνουμε είναι τα σωστά. Είναι φρόνιμο, κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη της Προεδρίας, να περιμένουμε, να δούμε από την Κομισιόν της θα μας δώσει στην αξιολόγηση τον Ιούνιο των μακροοικονομικών στρατηγικών. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό είναι ένα από τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση, που είναι το βασικό θέμα αυτής της Προεδρίας. Έχουμε πλήρη συνείδηση της σημασίας του θέματος. Αναφέρθηκε το θέμα της διασύνδεσης της Ευρώπης. Ήσασταν πολύ σύντομος, πολύ ακριβής και είπατε ότι έχετε ορισμένε ανησυχίε και νομίζω ότι θα μπορούμε να τις συζητήσετε. Να τις συζητήσουμε. Αναφέρατε και την εξοικονόμηση και αν αυτό μπορεί να διασυνδεθεί με το Ταμείο Συνοχής. Η Ιδανική Προεδρία θα το εξετάσει το θέμα αυτό με θετικό πνεύμα αλλά βεβαίως πολλές συζητήσεις θα πρέπει να λάβουν χώρα και χαίρομαι που υπάρχει ήδη ένας διάλογος με την Κομισιό για το θέμα αυτό, αλλά από την άποψη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της πράσινης ατζέντα που είναι το πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας και ε, είναι ευπρόσδεκτη κάθε πρωτοβουλία στο πλαίσιο αυτό. Μιλήσατε για το ρόλο των περιφερειών. Έχω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τις περιφέρειες και τις πόλεις επίσης. Εγώ είμαι πρώην δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Δανίας και ξέρω πολύ καλά ότι η χρήση κονδυλίων δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο από τους υπουργούς, γίνεται και επίση και σε τοπικό επίπεδο, με τρόπο επαγγελματικό. Και είναι αυτονόητο ότι οι περιφέρειες ως εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Και αυτό είναι και στην πρόταση της Κομισιόν και έτσι θα πρέπει να είναι. Και η Ιδανική Προεδρία θα ήθελε να συνεργαστεί με αυτή την Επιτροπή και με τις περιφέρειες για να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε σχετικά με το θέμα της αλληλεγγύης. Όπως ξέρετε, η ε, πρόταση της Κομισιόν του 2005 ε, προσέκλουσε σε αντίσταση από το Συμβούλιο, ξαναεξετάστηκε το 2006 στην ανακοίνωση του περασμένου Οκτωβρίου για το μέλλον του Ταμείου Αλληλεγγύης η Κομισιόν ανήγγειλε ότι τέλειψε την ιδέα της αναζωγόνησης πρότασης 2005. Απέσυρε την πρόταση. Αντίθετα, η Κομισιόν θέλει να εξετάσει τις δυνατότητες μιας νέας πρότασης που να τροποποιεί την, τον υφιστάμενο κανονισμό αργότερα. Και από ό,τι κατάλαβα, μια τέτοια πρόταση δεν θα υπάρξει κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας. Θα υπάρξει μόνο μια περιορισμένη προσπάθεια κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. θα ήθελα να κλείσω ε, μιλώντας δανέζικα, όπως είπατε, διότι δεν θέλω να απογοητεύσω τους διερμηνείς. Σας ευχαριστώ. Σε σχέση με αυτά τα θέματα θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς, σας, διερμηνείς μας ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης και γλώσσα τους και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την ευκαιρία που δίνεται τις απόψεις της Δανέζικης Προεδρίας να μπορέσουμε να τις παρουσιάσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν ευκαιρίες ε, όπου μπορεί να γίνεται αυτό. Ελπίζω ότι θα γίνονται όλο και πιο συχνές οι περιπτώσεις συμφωνίας. Αλλά υπάρχουν και διαφωνίες. Υπάρχει όμως η σαφέστατη πρόθεση της Δανέζικης Προεδρίας ότι θα θέλαμε με τέτοιο τρόπο να εργαστούμε ώστε με ανοιχτό τρόπο και ισοδίκαιο δίκαιο τρόπο να εργαζόμαστε με την Επιτροπή σας και με το Κοινοβούλιο τους Ευρωβουλευτές. Και χαίρομαι ήδη μπορώ να πω για τα αποτελέσματα Ελπίζω σύντομα με τους εισηγητές να μπορέσω να συναντηθώ σε αποστολή, για παράδειγμα με την Στην Κοπενχάγη είναι καλή προεδρία σε σχέση με τη Δανέζικη Προεδρία. Καλή πρωτοβουλία, με συγχωρείτε. Θα θέλουμε έτσι να σας καλωσορίσουμε, να σας υποδεχθούμε και το δυνατόν περισσότεροι σε αυτή τη διάσκεψη στην Κοπενχάγη να μπορέσουν να συμμετάσχουν όσον αφορά το MFR. Είναι μια τεράστια προ, ε, σημασίας πρωτοβουλία, μια πολύ καλή ευκαιρία, εξαιρετική ευκαιρία η Προεδρία, η Ευρωκοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη συζήτηση αυτών των θεμάτων σε, αυτές, σε αυτή τη σύνοδο, αλλά φυσικά και τα θέματα συνοχής ε, να συζητηθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα με αυτόν τον τρόπο για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα αυτή. Χαίρομαι ήδη ε, με την περαιτέρω συνεργασία που μπορούμε να έχουμε και για τις δικές σας προσπάθειες που καταβάλλονται και για το σαφές μήνυμα όλων, όλων που είπαν ότι από κοινού θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, να προοδεύσουμε προς των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω κύριε Υπουργέ, απλώς δύο λόγια. Θέλω να σας πω ότι εμείς αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή αναπτύξαμε την πραγματιστική προσέγγιση στο έργο μας που πρέπει να επιτελέσουμε Έχουμε δύσκολη χρονική συγκυρία και για μας το Ευρωκοινοβούλιο και για το Συμβούλιο και για, το Συμβούλιο, ε, και για την Επιτροπή. Είναι σημαντικό σταυροδρόμι αυτό τώρα στο οποίο βρισκόμαστε μπροστά για να λάβουμε τις αναγκαίες αποφάσεις. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ε, σε σχέση με τα όσα επιτελούνται στο Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε κάθε είδους συνεργασία, συναντήσεις ε, σε άτυπο και επίσημο επίπεδο και όχι μόνο επιτρέπετε να προσέλθετε, είσαστε ευπρόσδεκτο να προσέλθετε οποτεδήποτε θεωρείτε ότι έχετε κάποιε πληροφορίε που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μα να μα τι γνωστοποιήσετε. Ελπίζω ότι και από πλευρά του Στέφαν και τη συνεργασία που υπήρξε με την Τρόικα ότι θα μπορέσετε να συνεχίσετε να παρίσταστε και μέσα στο πλαίσιο των συμβουλίων, δύο γενικών συμβουλίων, γενικών υποθέσεων που θα γίνουν όπου θα εξεταστούν τα θέματα συνοχή. ελπίζουμε αμφωτέρωθεν και από τι δύο πλευρέ να διασφαλιστεί ότι αυτή η συνάντηση με το Ευρωκοινοβούλιο θα γίνεται όχι μόνο με του αρμόδιου για τα θέματα τα δημοσιονομικά, για τον προπολογισμό, αλλά και για, με του υπεύθυνου για τη χρηματοδότηση των θεμάτων για την πολιτική συνοχή, για παράδειγμα. Ένα από αυτά τα πεδία όπου εμεί θα θέλαμε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε ενεργά και από πλευρά μα. Αυτό θα ήθελα να ζητήσω να γίνει, να διασφαλιστεί λοιπόν ότι θα γίνει και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε να προσβλέψουμε στη μελλοντική συνεργασία με αυτό το πνεύμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ειλικρινή συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση με ειλικρινές πνεύμα που είχατε μαζί μας και για το σημερισμό, αν όχι όλων των απόψεων βέβαια, γιατί υπάρχουν φυσικά διαφορετικές απόψεις, όπως μπορώ να φανταστώ στο Συμβούλιο, δεν κάνω λόγο για τη Δανία, αλλά κάνω λόγο για την βούληση και την εμπλοκή και την ε, βούληση να σημειωθούν αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συνεδρίασή μας δεν ολοκληρώθηκε, δεν έληξε ακόμα, συνεχίζουμε. Παρακαλώ να παραμείνετε στην αίθουσα αν θέλετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συνεχίσουμε την συνεδρίαση. Τελείωσε το διάλειμμα, ας κάνουμε μια νέα κίνηση. Πρέπει επίσης να συνεχίσουμε και τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει πρωτού προσέθει ο υπουργό. Η συζήτηση για τον επιμερισμό δηλαδή των κινδύνων, το μέσο αυτό και τις τροπολογίες στον κοινό κανονισμό 2017-2013. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρίσταται. Εκπροσωπείται με τον Διευθυντή Βίσλερ. Έτσι, εσείς είσαστε. Υπάρχουν και άλλοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και την Task Force για την Ελλάδα ε, που εκπροσωπείται από τον κύριο Ράιχενμπα που θα παραστεί αύριο και που είναι επικεφαλής της Task Force ε, για την Ελλάδα Επίσης ε, και από τη Γενική Διεύθυνση έχουμε την κυρία Αντώνη. Όπως σας είπα πιο πριν, δεν ξεκινάμε από μηδενικό επίπεδο με αυτό το μέσο. Υπάρχει ήδη πείρα που έχει συσσωρευτεί, πραγματογνωμοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από προηγούμενα έτη, όπου διευκολύνσεις για τον επιμερισμό κινδύνου λειτουργήσαν. Έχουμε επίσης και την ιδέα, συγγνώμη, ε, και σε σχέση με την συμμετοχή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, από πλευράς Κριανκούν και για την ανταλλαγή απόψεων πριν από την συνάντηση με την Δανέζικη Προεδρία που είχαμε δύο πράγματα κυρίως ε, απορρέων και καθίστανται σαφή από αυτή τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που είχαμε σε αυτή την αίθουσα από την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Το θέμα του κατεπήγοντος πρώτον που πιέζει 2012-2013. Έχουμε δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που πρέπει να χρησιμοποιηθούν με δραστήριο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε με αυτό το μέσο. Δεν υπάρχει πολλής χρόνος, υπάρχει κατεπήγον χαρακτήρας. Πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα, να σημειωθεί ανάπτυξη, να υπάρξει ανάπτυξη για τις οικονομίες των χωρών αυτών που εμπλέκονται. Και γι' αυτό ανησυχούμε κάπως πρέπει να πω, σε σχέση και με αυτά που επιβεβαίωσε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ότι δεν έχει δηλαδή κινηθεί ακόμα, κινητοποιηθεί το Συμβούλιο. Και σε σχέση με την τεχνική ενημέρωση που θα έχουμε αύριο, ελπίζω ότι θα υπάρχει αλλάξει το εναρκτήριο λάκτισμα, θα, θα δώσουμε τον εναρκτήριο πυροβολισμό για να ξεκινήσουν όλα αυτά. Τώρα και από την ανταλλαγή απόψεων για, αυτά, για αυτό το μέσο είναι πολύ σημαντικές κάποιες πτυχές, θα έλεγα ζωτική σημασίας, παρότι αφορούν την κάλυψη γεωγραφικά όσο αφορά την επικράτεια, αλλά και την επιλεξιμότητα σχεδίων. Η επικρατούσα άποψη στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή ποια είναι είναι ότι εμείς ως ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή θεωρούμε ότι η στόχευση, η επικέντρωση θα πρέπει να είναι στα θέματα πολιτικής συνοχής. Πολλά επιχειρήματα ακούγονται και διατυπώθηκαν, αλλά αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα θέλαμε να, να ακούσουμε από εσά τώρα τα επιχειρήματα υπέρ της διεύρυνσης ή μη διεύρυνσης, μη επέκτασης των δυνατοτήτων επιλεξιμότητας σχεδίων όσον αφορά τις προτάσεις που έχουν τεθεί για την πολιτική συνοχή ή και πέρα από αυτήν. Δεύτερο θέμα το οποίο αφορά αυτή την κάλυψη είναι το γεωγραφικό ζήτημα της γεωγραφικής κάλυψης επικράτειας γεωγραφικά. Ανοίγει το ερώτημα εδώ. Αυτό δεν θα προσέθεται πολύ στο βάρος που θα υπομιζόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτό το μέσο. Αν δεν περιοριστεί γεωγραφικά στα έξι κράτη-μέλη αυτό το μέσο σε σχέση με την προηγούμενη τροποποίηση του κανονισμού για την δράση με αυτά τα κονδύλια. Αυτά τα θέματα απομένουν. Όλα τα άλλα τεχνικά θέματα, εκτός αν κάποιος ε, τα αναφέρει ξεχωριστά, με την τεχνική ε, υφής ενημέρωσης που, ενημέρωση που είχαμε πριν από δύο εβδομάδες θεωρούμε ότι ήταν με χρήσιμο τρόπο μπόρεσαν να διευθετηθούν και να συμφωνηθούν. Αν μπορείτε τώρα λοιπόν να επικεντρωθείτε σε αυτά τα επιχειρήματα υπέρ ή κατά Τη επέκταση, τη διεύρυνση τη επιλεξιμότητα και υπέρ ή κατά τη διεύρυνση τη επέκταση τη γεωγραφική κάλυψη ω κριτηρίου. Διότι αυτό θα ήταν χρήσιμο. Και όπως ξέρετε, σε σχέση με την ε, ομάδα εργασίας Task Force για την Ελλάδα, που εχθές στην Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών ε, συζήτησε κάποια θέματα, είχαμε και το θέμα της γνωμοδότησης και υπέρ, έκφρασης, ε, υπέρ της επέκτασης της εμβέλειας της δράσης αυτού του μέσου. Αυτό πληροφοριακά μόνο σα το αναφέρω. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Ρούντολφ, νομίζω πρώτα. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πολλά ευχαριστώ στη συνέχεια για το ότι διοργανώσατε αυτή την τεχνική συνάντηση όπου θεωρούμε ότι έχουμε μια ευκαιρία να εξετάσουμε ένα σημαντικό εύρος ζητημάτων για την επιλεξιμότητα, για παράδειγμα, για την λειτουργία και λειτουργικότητα του μέσου και για το να συμμεριστούμε τις πύρα, την πείρα, τις εμπειρίες των συναδέλφων που παρήσατε σήμερα ανάμεσά μας για το τι πραγματικά συμβαίνει στο πεδίο επιτόπου. Και έχουμε και τους συναδέλφους και τον κύριο Ράιχενμπαχ ιδιαίτερα που παρίστανται, που θα μπορέσουν να επεξηγήσουν πώς έχει η τελευταία φάση όλων αυτών των δράσεων συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Θα ήθελα να στραφώ στο ερώτημά σα τώρα άμεσα στη συνέχεια Πρόεδρε. Πριν το κάνω αυτό να πω ένα πράγμα μόνο. Η πρόταση όπω γνωρίζετε εμπνεόταν από την συγκεκριμένη κατάσταση όπω είχε διαμορφωθεί και την οποία αντιμετωπίσαμε στην Ελλάδα. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε στην Ελλάδα. Απειλή σε μεγάλο βαθμό των δράσεων ε, όσον αφορά τις δράσεις στον τομέα των υποδομών που έπρεπε να διασφαλιστούν όπου ε, είχαμε θέματα χρηματοδότησης, συγχρηματοδότησης και επειδή υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα υπάρχουν προβλήματα στον τραπεζικό τομέα να συνεισφέρει στην ε, ρευστότητα και η συνεισφορά από πλευρά των εταίρων αυτών των σχεδίων οικονομικά δεν μπορούσαν να προαχθούν και αυτά τα σχέδια και προγράμματα είχαν σταματήσει πλέον δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν είναι σημαντικό για μας να διασφαλίσουμε λοιπόν τα μέτρα αυτά, τα μέσα για την πολιτική συνοχή σε αυτόν τον πολύ σημαντικό τομέα και να μεριμνήσουμε και να διασφαλίσουμε και αυτό το θέμα της πρόσθετης χρηματοδότησης ε, που θα έπρεπε να δοθεί σε αυτά τα σχέδια. Αυτή είναι, ας το έτσι, αυτό είναι το ένασμα, η προέλευση αυτής της πρότασης που από κοινού αναπτύξαμε και διατυπώσαμε με τους συναδέρφους μας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το ΕΚΟΦΗΝ η γραμμή αφετηρίας είναι λοιπόν η αντιμετώπιση της κρίσης με συγκεκριμένες δράσεις και διασφάλιση του συντονισμού των σχεδίων και μέτρων προγραμμάτων για την συνοχή. Υπό το δικό μας πρίσμα, στρεφόμενος τώρα στα συγκεκριμένα ερωτήματα που διατυπώσατε Πρόεδρε, αν θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την διεύρυνση της εμβέλειας του φάσματος αυτής της πρότασης σε ένα μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως αντιμετώπιση της κρίσης αυτό το μέτρο. Και εμείς πιστεύουμε ότι η άποψή μας για να είμαστε συνεπείς πρέπει να είναι ότι θα περιορίζεται αυτό το μέσο σε εκείνες τις χώρες για τις οποίες είχαν ήδη προταθεί και με τροπολογίες συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθηθούν αυτές οι χώρες ευθυγραμμίζεται αυτό και συνεχίζει την ίδια κατεύθυνση όπως για την άλλη πρόταση, δηλαδή αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης από πλευράς μας, που συμφωνήθηκε αυτό πέρυσι να αυξηθεί το επίπεδο ε, χρηματοδότησης από εμάς. Από ό,τι ε, είναι σαφές ε, δεν πρόκειται για κάποιον αυτοματισμό αυτού, δηλαδή για τον επιμερισμό των, ε, των κινδύνων σε αυτές τις έξι χώρες ε, υπό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Σαφώς λοιπόν αναφέρεται ότι μόνο με αίτημα των κρατών μελών θα γίνεται αυτό. Δηλαδή με βάση μια προσεκτική ενδελεχή ε, ανάλυση ε, ανακράτος και αναδράση, ανασχέδιο αν θα πρέπει να γίνει αυτό ή όχι. Αυτό για τις έξι αυτές χώρες, για τις δράσεις που θα ακολουθηθούν αποτελεί λιδία λίθο. Όπως έχουν τα πράγματα τώρα, δεν έχουμε λάβει μηνύματα από άλλες χώρες πέρα από τις έξι αυτές που να λένε ότι θα θεωρεί το αναγκαίο ή κατεπήγον να επεκταθεί αυτή η δράση σε εκείνα τα κράτη σε αυτή τη φάση. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι η επικέντρωση θα πρέπει να είναι στην αντιμετώπιση της κρίσης σε έκτακτα μέτρα, ειδικά μέτρα και λαμβάνοντας υπόψη αυτέ τις ακραίε καταστάσεις που δημιουργούνται και που διακυβεύουν την ε, ανάπτυξη και την εξέλιξη των ε, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σχεδίων σε σχέση με αυτές τις χώρες. Πρέπει να, να έχετε συνειδητοποιήσει ότι και για αυτές τις χώρες στις οποίες στοχοθετούμε σε αυτή την πρώτη φάση δεν θα μπορούσε να προχωρήσει τίποτα αν μια χώρα έχανε τα κονδύλια της από την πολιτική συνοχή, επειδή δεν θα μπορούσε η χώρα αυτή να διεκδικήσει το ποσοστό εκείνο χρηματοδότησης που θα ήταν εφικτό να διατεθεί σε εκείνο το ε, σκέλος όπου υπάρχει η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί η δική της συγχρηματοδότηση. Η πρόταση λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ένα μέρος των μη διατεθειμένων κονδυλίων ώστε να χρησιμοποιηθούν τα μη αντληθέντα κονδύλια προς αυτές τις αρχές ώστε να απορροφηθούν ως ε, δαπάνες για, για την εξέλιξη αυτών των σχεδίων είναι σημαντικό μέτρο. Διαφορετικά θα έχαναν οι χώρες κονδύλια από αυτά τα ε, προγράμματα. Είναι στρατηγικού χαρακτήρα, στρατηγικής ευρωπαϊκής φύσης ε, ε, ως προς το χαρακτήρα αυτά τα μέτρα. Έχουμε και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικά πολύ σημαντικών ε, τέτοιων ε, προγραμμάτων και σχεδίων. Ο κύριος Ράχενμπαχ είμαι βέβαιος ότι θα επεκταθεί περισσότερο στη συνέχεια από αυτών. Δεύτερον, γιατί επικεντρωνόμαστε στην πολιτική συνοχής επίσης ή μόνο. Πώς συμβαίνει αυτό. Ο στόχος όπως το ανέφερα είναι να διασφαλιστεί η υλοποίηση της πολιτικής συνοχής όσον αφορά τη στρατηγική που είχαμε εκπονήσει. Και στην φάση υλοποίηση στην οποία βρισκόμαστε θα ήταν, δεν θα ήταν καθόλου ευκταίο να ε, διαλάθη να μπορέσει να αγνοηθεί η ανάπτυξη αυτών των σχεδίων που βρίσκονται υπό εξέλιξη αλλά έχουν διακοπεί λόγω της κατάστασης κρίσης. Ε, Εμεί θεωρούμε ότι η προτεραιότητα είναι να συνεχιστεί η εξέλιξη αυτών των σχεδίων και να δοθεί συνέχεια σε αυτά και να μην παρεκκλίνει, α το πω έτσι, η ενεργητικότητά μα και τα κονδύλια μα στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και σχεδίων που δεν θα υπήρχε βεβαιότητα ότι θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν και να υλοποιηθούν μέσα στα πλαίσια τη τρέχουσα περίοδου. Όλα αυτά βλέποντας ένα, με μια ματιά το χρονοδιάγραμμα αμέσως επεξηγούνται αφ' αυτόν. Έχουμε δύο χρόνια ακόμα για την υλοποίηση προγραμμάτων και σχεδίων σε αυτή την περίοδο προσεγγίζοντας αυτή την ε, καταληπτική ημερομηνία θα μπορούσαν τέτοιου είδους ε, προγράμματα που θα θέλαμε να ξεκινήσουν να ξεκινήσουν από το 2014 και εφ' Μέχρι τότε πρέπει να ολοκληρώσουμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά την επιλεξιμότητα τέτοιων σχεδίων. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής Πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες και κανονισμούς και εθνικούς κανόνες και κανονισμούς για την επιλεξιμότητα των δράσεών μας. Θα πρέπει να αποκλίνουμε, να παρεκκλίνουμε από αυτές τις αρχές. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, πολλά ερωτήματα θα έπρεπε να απαντηθούν. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν θα μπορούσε αυτό να στεφθεί με επιτυχία και αν θα συνεισέφερε επικοδομητικά μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης της εξέτασης αυτών των προτάσεων εδώ και εδώ και στο Συμβούλιο. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε αυτή την περίπλοκη ακαθόδη υπερβολικά σύνθετη συζήτηση του να εξετάσουμε μια διεύρυνση, μια επέκταση των κανόνων και κανονισμών πέρα από το πεδίο της πολιτικής συνοχής. Τούτων λεχθέντων, κυρία Πρόεδρε, επαρκούμε σε αυτά τα σχόλια. Αυτά ήθελα να πω με ευχαρίστηση ας συμπληρώσουν οι συνάδελφοι αν επιθυμούν. Ευχαριστώ. Very much, very... Ευχαριστώ πολύ. Ε, πολύ σύντομα δεν ξέρω αν ποιος θέλει ε, να λάβει τον λόγο. Είστε πρόσδεκτος. Ίσως απλώς να πω ότι αυτά τα οποία αναφέρατε στην αρχή το κατεπήγοντα χαρακτήρα παραμπτός χάρη είναι κάτι το πολύ σημαντικό για την Ελλάδα κυρίως για τα έργα, οι παραχωρήσεις, οι εκχωρήσεις που έχουν γίνει για αυτοκινητοδρόμους, παραμπτός χάρη. Είναι λοιπόν κατεπήγον το μέτρο αυτό. Θα πρέπει τα τέσσερα έργα τα οποία δεν προχωρούν καλά με ικανοποιητικό τρόπο να μπορέσουν να επιταχυνθούν όσον αφορά ε, την ε, πολιτική συνοχή, η οποία είναι η πρώτη προτεραιότητα στην Ελλάδα από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπαδήμο. Γίνεται, γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε αυτό να καταστεί εφικτό. Ακόμα και χωρίς αλλαγή στον κανονισμό αλλά χωρίς αλλαγή στον κανονισμό υπάρχει πολύ λίγη ελπίδα να περατωθούν αυτά τα έργα. Και θα σας πω γιατί είναι τόσο σημαντικό από χρηματοοικονομικής απόψεως, όχι μόνο από την άποψη της συνοχής, αλλά επίσης και από της ελληνικής πλευράς. Διότι εάν τα έργα αυτά δεν συνεχιστούν, ε, τότε αυτοί που έχουν την εκχώρηση, που έχουν ε, συμβάσεις, ε, θα έχουν απαιτήσει και αυτές οι απαιτήσει μπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλέ. Δεν είναι λοιπόν θέμα να αρχίσουν αυτά τα έργα, είναι θέμα να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα για να αποφευθούν αυτές οι απαιτήσει εκ μέρους των δικαιούχων ε, των εκχωρήσεων. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα έργα τα οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν από το μέσο επιμερισμού του κινδύνου, αλλά νομίζω ότι τα έργα οδοποιίας στην Ελλάδα έχουν πάρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, ε, υπάρχουν και άλλες παρατηρήσεις. Ναι, είμαι από τη DG Ekfield. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα που λέχτηκαν τελευταία φορά στην τεχνική συνάντηση. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Το μέσο υπάρχει εδώ και έξι χρόνια για τα έργα υποδομών, για τις έρευνες και συνεπώς ε, βασιζόμαστε σε κάτι που υπάρχει που είναι ένα μέσο διαφανέσα υποστήριξης των υποδομών. Όλα τα προγράμματα και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τα έργα τα οποία ωφελήθηκαν από αυτή τη χρηματοδότηση δημοσιεύοντα. Αναφέρουμε στην αρχή του προϋπολογισμού για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες διαθέσιμες και αυτό νομίζω ότι απαντά στις ερωτήσεις αν υπάρχουν και είμαστε και εμείς στη διάθεσή για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που έχω να πω μερικά λόγια για αυτήν την εξαίρετη πρωτοβουλία για την οποία ευχαριστούμε την Κομισιόν που έκανε την πρόταση. Έχουμε δύο σημεία τα οποία αναφέρατε εσείς στην αρχή και θέσατε επιτάπητος. Πρώτα απ' όλα τον κατεπήγοντα χαρακτήρο του θέματος. Νομίζω ότι ο κανόνας του παιχνιδιού και όχι μόνο ε, κατεπήγουσα η απόφαση αλλά κατεπήγουσα και η υλοποίηση της απόφασης. Εάν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα εφαρμόσουμε, θα υλοποιήσουμε την απόφαση, είναι πολύ σημαντικό οι προϋποθέσεις, οι όροι που θα τεθούν να επιτρέπουν μια ταχύτατη υλοποίηση. Γι' αυτό νομίζω ότι το θέμα της επιλεξιμότητας πρέπει να εξεταστεί πάρα πολύ προσεκτικά ε, διότι τα λειτουργικά επιχειρησιακά προγράμματα αποφασίστηκαν σε διαφορετικό χρόνο η κρίση και οι προτεραιότητες ίσως έχουν αλλάξει σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένες χώρες και σε ορισμένες καταστάσεις. Μερικά έργα έχουν μπλοκαριστεί και γι' αυτό τα διαρθρωτικά ταμεία δεν έχουν ξοδευτεί τα κονδύλια τους, αν έχουν μπλοκαριστεί, ίσως υπάρχουν ε, προβλήματα με τα ίδια τα έργα αυτά και θα μπορούσαν άλλα έργα, ακολουθώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προτεραιότητες, θα μπορούσαν να αναλάβουν τα, το έργο αυτό με τα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής. Η ευελιξία, συνεπώς, είναι σημαντική. Η απόφαση που λήφθηκε και που είναι καλή για την αύξηση του μέγιστου ε, ποσοστού μέχρι 95% που θα ε, επιδοτείται, νομίζω είναι ένα άλλο μέσο, διότι εάν ε, το όλο ε, μέσο καλύψει 5% ίσως δεν επιτυγχάνουμε το στόχο μας. Ίσως θα πρέπει να ανοίξουμε το, την πόρτα για άλλα έργα που απαιτούν περισσότερα, περισσότερη χρηματοδότηση. Ξέρουμε ότι για όλους αυτούς τους λόγους ε, έχουμε την, ε, τη διαδικασία αυτή η οποία όπως αναφέρθηκε είναι διαφανής, ελεγχόμενη, αναφερόμενη. Θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί πλήρως ε, ούτω ώστε να υπάρξει η υλοποίηση ταχύτατα μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα πριν από τις προθεσμίες. Αυτό για το θέμα της επιλεξικότητας ε, και ε, βεβαίως χωρίς να θίγονται οι προτεραιότητες όπως αυτές ε, που μας ανέφερε ο κύριος Ράιχεμπαχ των αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα είναι ένα μήνυμα που καταλαβαίνουμε πλήρως αλλά και η ευελιξία είναι για μας σημαντικό θέμα ως προς τις χώρες και την γεωγραφική κάλυψη. Η κρίση είναι το βασικό κριτήριο, όπως λέχθηκε. Νομίζω ότι η κρίση υπερβαίνει τα όρια των χωρών του προγράμματος. Υπάρχουν μερικές μεγάλες χώρες οι οποίες βρίσκονται επίσης σε κατάσταση κρίσης. Αν χρειάζεται χρόνος για να αλλάξει ο κανονισμός, αν δεν υπάρχει ανακατανομή κλπ. και αν η δικαιούχος χώρα που πρέπει να αποφασίσει για τη χρήση για το μέσον ε, δεν ε, αποφασίζει, δεν βλέπω γιατί να διευρυνθεί σε άλλες χώρες. Αλλά πρέπει να επανέλθουμε σε όλη την ε, κανονιστική άσκηση και αν σε έξι μήνες θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Ίσως σήμερα θα είναι εσφαλμένη η απόφαση να περιορίσουμε σε αυτές τις χώρες. Δεν είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε, είμαστε εδώ για να ακούσουμε τα επιχειρήματα ε, δεν ε, είσαστε πολύ χρήσιμοι για τις αποφάσεις ε, για αυτήν την Επιτροπή. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω μια διευκρίνηση σε αυτά που είπα, λέχθηκαν. Δεν είναι το 5% που θα εξασφαλιστεί από το μέσο. Το 5% που ανέφερε η Ντομινίκ θα είναι η συναχρηματοδότηση. Ε, που είναι μέσα στο, στην χρηματοδοτούμενη τρύπα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ε, το θέμα είναι τι δεν καλύπτεται η συμβολή του ιδιωτικού ε, τομέα που έχουμε σε αυτές, αυτά τα σχέδια εκχωρήσεως. Αυτά είναι τα τμήματα των έργων που δεν καλύπτονται, δεν εξασφαλίζονται στις αυτοκινητοδρόμους της Ελλάδας, για να σας δώσω μια ιδέα. 50% του συνολικού κόστους καλύπτεται από ε, την χρηματοδότηση ε, την ευρωπαϊκή 95% και 5% προέρχεται από την εθνική συγχρηματοδότηση, αλλά υπάρχει και ένα ίσο ποσό που προέρχεται από τους άλλους συνεισφέροντες στο έργο. Αυτό είναι όγκος της χρηματοδότησης που θέλουμε να καλυφθεί. Μικρόφωνο παρακαλώ, νομίζω χωρίς μικρόφωνο παρέμβαση. Με συγχωρείτε. Ε, διαρωτώ ε, με αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από μάσα. Εάν όχι, νομίζω τότε ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης Ελπίζω ότι θα έχουμε την έκθεση για ε, την επόμενη ε, συνεδρίαση. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω ότι το θέμα είναι κατεπήγον και θα πρέπει να ακούσουμε και άλλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Task Force για την Ελλάδα. Κλείνω με το θέμα και τώρα έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Όλοι οι άλλοι παρακαλούνται να φύγουν από την αίθουσα και να μείνουν μόνο οι συντονιστές.